Colleagues, Μήπως μπορείτε να καθίσετε κύριοι συνάδελφοι γιατί θέλω να αρχίσω. Θέλω να αρχίσω. Έχουμε στην αρχή το τέλος της Ρέγγι του πρωινού Έχουμε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης της Πολωνίας και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Τσεχίας, Δανιήλ Μπράουν. Ίσως πρώτα ο πιο υψηλόβαθμος. Πρώτα την Πολωνία θα ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Καθηγήτρια Χιούμπνερ, κυρίες και κύριοι, λίγοι πιστεύουν ότι σύντομα θα πετύχει η πολιτική συνοχή της Ένωσης εύκολα ή σύντομα και ιδίω οι χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πολλά προβλήματα παραμένουν εκκρεμή με διαθροτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν πολύ σύντομα. Θα μπορέσει όμως η κυβέρνηση των χωρών αυτών, όλων των χωρών να εφαρμόσει αυτό το νέο σύστημα επιτυχώς. Και τέλος, οι εθνικοί προϋπολογισμοί θα μπορέσουν να φέρουν το βάρος της χρηματοδότησης. Σήμερα ξέρουμε ότι καταφέραμε στην Πολωνία να γίνουμε ο μεγαλύτερος αποδέκτης κονδυλίων για την περιφερειακή ανάπτυξη και υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα της χρήσης των κοινοτικών ταμείων. Από τα κύρια αποτελέσματα είναι η εφαρμογή της μεγαλύτερης ανάπτυξης εξυγχρονισμού στην πολωνική ιστορία ολόκληρη που χρησιμοποιήθηκε ως ε, αφετηρία για περισσότερη ανάπτυξη και περιορισμό των ε, ζημιών από εξωτερικές συνθήκες για τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών. Η δε ανάγκη να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής αναγκάσε την πολωνική κυβέρνηση σε διαφορετικά επίπεδα να εφαρμόσει τις αλλαγές που είναι απαραίτητες για να είναι πιο αποτελεσματική και άρα ενδυνάμωσε τη δυνατότητά της σχεδιασμού. Όλα αυτά κατέληξαν σε μια επιταχυμένη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σημαντική μείωση του χάσματος μεταξύ Πολωνίας και των πιο ανεπτυγμένων χωρών της Ένωσης και ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Στην Πολωνία η πολιτική συνοχή σημαίνει ανάπτυξη. Μεταξύ του 7 και του 12 η πολωνική οικονομία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 4% σε σύγκριση με το μέσο όρο του 0,2% στην Ένωση. Εκτός αυτού συνεχίσαμε στον δρόμο αυτό ακόμη και κατά τα χρόνια της χρήσης 9 με 10 λόγω της υψηλής, του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ 7 με 12, το χάσμα μεταξύ Πολωνίας και των 20, του μέσου όρου των 27 της Ένωσης ως ε, κατακεφαλήνα ΕΠ ή ως αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί κατά 14 εκατοστιαίες μονάδες. Λόγω δε του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης οι συγκλήσεις σημείωσαν ότι η Πολωνία ήταν η πρώτη σε αυτό το θέμα και αναμένουμε να καταλήξει σε ρυθμό 70% να καλύψει το 70% του κοινοτικού κεκτημένου και αυτό θα οφείλεται εμπολής στα ενωσιακά κονδύλια. Αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα διότι το 12 πέρυσι δηλαδή είχαμε φτάσει μόνο στο 66%. Οι θετικές λοιπόν επιπτώσεις της ε, πολιτικής συνοχής της Ένωσης φαίνονται σε πολλούς τομείς. Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, μεγαλύτερη κατάρτιση και καλύτερη κατάρτιση των εργαζομένων και συνθήκες εργασίας, εξυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών και μεταξύ των οποίων και η οικοδόμηση αυτοκινητοδρόμων που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη συνοχή της Ευρώπης. Και αυτά όλα είναι αδιαμφισβήτητα. Οι επιχειρηματίες επωφελήθηκαν από τη στήριξη των κοινοτικών κονδυλίων και από τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Και τώρα είναι ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά όχι μόνο λόγω της χαμηλότερου κόστους παραγωγής αλλά κυρίως λόγω των καινοτόμων προϊόντων που παράγουν. Για να συνοψίσω, τα ενωσιακά κονδύλια επέτρεψαν στην πολωνική οικονομία να γίνει πιο καινοτόμα και πιο ανταγωνιστική και έτσι να ανταποκρίνεται πιο εύκολα στις νέα, στο νέο είδος ζήτησης. Οι υποδομές, και η άμεση στήριξη στις επιχειρήσεις με κοινοτική επιχορήγηση οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά 20-25%. Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν μετά από την εφαρμογή των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση υπολογίζεται σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδων. Εκτός αυτού η Πολωνία είναι χώρα όπου καταγράφηκε μετά τη Γερμανία η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας την περίοδο 7 με 12 κατά 3,8%. Due... Αυτό δεν πολύ οφείλεται στη χρήση των κοινοτικών κοντιλίων αλλά ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η πολιτική συνοχή εργάζεται με δύο τρόπους δηλαδή έχει και σχετίζεται και με τις υπόλοιπες χώρες. Τα ερευνητικά ιδρύματα υπολόγισαν τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής για το λεγόμενο EU15 ως ε, επιστροφή κέρδος 61 λεπτών ανά ευρώ με τη μορφή πρόσθετων εξαγωγών, συμβολέων και επιχορηγήσεων. Η σχετική μελέτη δείχνει ότι η πολιτική συνοχή λοιπόν μεταξύ άλλων βελτιώνει το σύνολο της Ένωσης και συνεισφέρει και στην περιφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη που με τη σειρά της προωθεί το εμπόριο και την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο και σταθεροποιεί την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την περιφερειακή συνοχή. Η πολωνική εμπειρία 7 με 13 στις δημοσιονομικές προοπτικές δηλαδή δεν είναι όμως μόνο θετική γιατί χρειάστηκε να καταπολεμήσουμε και τις ελλείψεις του συστήματος που οφείλονται κυρίως σε ασαφείς διευθετήσεις που απαιτούν συνεχή ερμηνεία από την Κομισιόν και πολλές φορές υπάρχουν παρεξηγήσεις από τους δημοσιονομικούς ελεγκτές. Επιβάλλονται άχρηστα διοικητικά βάρη και άχθη για να εγκριθεί οτιδήποτε από την Κομισιόν. Όλα αυτά όθησαν στην ε, έγκριση αλλαγών για την επόμενη περίοδο. Μηχανισμούς δηλαδή για περισσότερη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, πράγμα που φαίνεται από ενισχυμένη συνεργασία των ε, δημοσιονομικών εργαλείων και οργάνων της Ένωσης, θεματική συγκέντρωση και προσέγγιση που να βασίζεται στα αποτελέσματα. Η Πολωνία συμμετέσχε στη διατύπωση των αναπτυξιακών προτάσεων στην Ένωση και χαίρομαι γιατί καταφέραμε να δεχτούμε λύσεις απλοποίησης της εφαρμογής της χρήσης των κοινοτικών κονδυλίων. Διότι η δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου συστήματος είναι το μισό, είναι το μισό πρόβλημα Μεταξύ άλλων μέτρων είναι οι κοινοί κανονισμοί για τη χρήση των πέντε ταμείων και άρα απλοποιημένη χρήση και υπολείπων όπως του αλλιευτικού. Έτσι αυξάνονται και τα κατώτατα όρια για την εφαρμογή διαφόρων σχεδίων και ψηφο, ψηφιοποιούνται όλα αυτά. Αυτές οι αλλαγές σίγουρα θα έχουν θετικές επιπτώσεις και για τους ανθρώπους και για τους οργανισμούς που ασχολούνται με την πολιτική συνοχή. Και με αυτή την ευκαιρία ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία μας στις διαπραγματεύσεις ως προς το νομο, την νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχή που σε λίγο θα καταλήξει. Η συνεργασία με την Επιτροπή Περίφ συγκεκριμένα είναι υποδειγματικοί. Έχουν γίνει πάρα πολύ καλές συζητήσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο και για άλλες επιτροπές. Μερικά θέματα ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας δεν έχουν ακόμα λυθεί πριν λήξουν οι διαπραγματεύσεις με τους ε, τριμερείς διαλόγους και αφορούν κυρίως τη δημοσιονομική διαχείριση μακροοικονομική αιρεσιμότητα και την πρωτοβουλία απασχολησιμότητας των νέων. Αυτά είναι δύσκολα και πολύπλοκα θέματα, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε καμία λύση που θα παρέλειε την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και θα μείωνε την αποτελεσματικότητά της. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω μερικές σκέψεις μου για το πώς θα μπορούσε να προφευχθεί μια τέτοια αρνητική κατάσταση. Καταρχήν η μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Θέμα που έχει δημιουργήσει μεγάλες διαμάχες και διαφωνίες και η τελευταία θέση του Συμβουλίου αποδείχθηκε δύσκολα διαπραγματεύσιμη. Για την Πολωνία οι δυσκολίες αυτές δείχνουν ότι πρέπει τα όργανα να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να εγκριθούν διαδικασίες που να αποφεύγουν τις πολλαπλές και αντιμαχόμενες ερμηνείες. γνωρίζουμε την ανάγκη να ενδυναμωθεί η λειτουργία των οργάνων διακυβέρνησης, οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση ώστε να υπάρξουν σταθερές και βιώσιμες μακροοικονομικές συνθήκες για να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής του 2020. Και αυτόν τον λόγο πιστεύουμε ότι η μακροοικονομική ρεσιμότητα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Εάν η μακροοικονομική ρεσιμότητα εφαρμοζόταν μόνο στο Ταμείο Συνοχής όπως γίνεται τώρα, τότε θα αφορούσε μόνο τις χώρες που ωφελούνται από το Ταμείο αυτό. Και έτσι θα δημιουργηθεί ένα αίσθημα αδικίας. Χρειάζεται φρόνηση για τον καθορισμό των σχέσεων μεταξύ οικονομικής διακυβέρνησης και χρήσης των ενωσιακών ταμείων. Η μικροοικονομική αιρεσιμότητα δεν είναι δυνατόν να παραλύσει τη λειτουργία των ταμείων και δεν πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαιότητας ως προς τις προσδοκίες που αναμένουν τα κράτη-μέλη. Επίσης σημαντικό είναι να διασφαλιστεί μια πραγματική, πραγματιστική σχέση μεταξύ όλων αυτών. Από την άποψη της Πολωνίας, η σχέση αυτή είναι αφισβητήσιμη. Άλλο θέμα είναι το πλαίσιο αποτελεσματικότητας performance framework θεωρούμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος χρηματιασμός και εφαρμογή του. Και αυτό το βασίζουμε στην τωρινή προγραμματική περίοδο. Η Πολωνία είναι μία από τα δύο κράτη-μέλη που έχουν εφαρμόσει το αποθεματικό αποτελεσματικότητας πιο σοβαρά από όλες τις χώρες. Και λόγω των σημαντικών πολιτικών επιπτώσεων που έχει αυτό το performance framework δεν πρέπει να υπάρξει καμία ασάφεια νομικά ως προς τις συνθήκες που το διέπουν. Το εργαλείο αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να λάβουμε υπόψη μας και την τρέχουσα την τωρινή κατάσταση και το γεγονός ότι πρέπει να βελτιωθούν οι μέθοδοι καθορισμού των στόχων και των μέτρων με τους οποίους θα επιτευχθούν. Άλλη παρατήρηση ως προς την δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες για να μην υπάρχει σύγχυση. Και γι' αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό τον καθορισμό της ενίας της ατασταλίας και της συστηματικής ατασταλίας και να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα κριθεί αυτό. Καταλήγοντας ελπίζω ότι οι εμπειρίες και προτάσεις της Πολωνίας και άλλων που ωφελούνται από την ε, πολιτική συνοχή θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής στο σύνολό της στο μέλλον και προσβλέπω σε σύντομη κατάληξη των διαπραγματεύσεων ως προς την πολιτική συνοχή ε, την, δέσμη δηλαδή για να υπάρξει καλύτερη χρήση ήδη από την αρχή του 2014 των αναπτυξιακών ταμείων που πιστεύω ότι είναι ο κοινός μας στόχος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, um, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κούμπιακ. Συνήθως δεν χειροκροτούμε. Δείχνει αυτό πόσο εξαιρετική ήταν η παρουσία σας. Παρακαλώ τώρα τον επόμενο μιλητή, τον, τον κύριο Μπράουν, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μου ζητήθηκε να δώσω τις δικές μας τοποθετήσεις και την κριτική θεώρηση τόσο από τη δική μας πλευρά όσο και κοιτώντας προς τα έξω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο έχει ένα πολύ ισχυρό ρόλο για την βελτίωση και την ενίσχυση της αντίληψης του πώς λειτουργούν η περιφερειακή πολιτική και τα διαφορετικά ταμεία. Θα ήθελα να δώσω μια σύντομη συνεισφορά από πλευρά μου προς την, για την ευρωπαϊκή πολιτική που αποτελεί απτή ένδειξη αλληλεγγύης μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών και πολιτών. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ από πλευρά της δημοκρατίας, δημοκρατίας στην, ε, στην εμπειρία μας με, το θετικό αντίκτυπο. Δεύτερον, να αναφερθώ στα διδάγματα της επόδυνης μερικές φορές διαδικασίας. Και τρίτον, να στραφώ στο μέλλον και την ε, προβολή σε μελλοντικά προγράμματα. Θα αναφερθώ επίσης τέταρτον στους εξωγενείς παράγοντες που έχουμε εντοπίσει για το τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα και στο μέλλον σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή και πολιτική, η οποία θα επιτρέπει την ανάπτυξη των περιφερειών και όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν συνεχίσουμε να μεγιστοποιούμε την, την αποτελεσματική χρήση των πόρων που διατίθενται. Και ξεκινώ λέγοντας ότι είναι μια ε, μεσαία, μεσαίου μεγέθους χώρα η Τσεχία, κεντρική ε, χώρα στην κεντρική Ευρώπη, 10 περίπου εκατομμύρια κατοίκους. Ξέρετε ότι το 2004 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως τώρα διανύουμε την πλήρη προγραμματική περίοδο. Η πρώτη που ήταν σύντομη, 2004-2006, αξιοποίησε μέσω των τσεχικών προγραμμάτων περίπου 2,6 δις ευρώ, ενώ στην τρέχουσα έχουμε στη θέση μας 26,7 δις ευρώ, 60 περίπου τις 100 εκ των οποίων έχουν ήδη καταβληθεί στον τελικό δικαιούχο. Η τσεχική δημοκρατία επίσης είναι μια οικονομία ανοιχτή με 80 περίπου τις 100 του ΑΕΠ κατά μέσον όρο και κατά κεφαλήν. Έχουμε, όπως και στα πολλά άλλα κράτη-μέλη βεβαίως, μια περιοχή πρωτεύουσα που παρουσιάζει πολύ διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια και θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν ε, προβλήματα υπανάπτυξης υποδομών και υποστήριξης, αναγκαίας υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που αξιοποίησαν κατά πολύ χρήσιμο τρόπο οι τοπικές αρχές, περιφέρειες, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είμαστε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της περιοχής μας ως προς τα χαρακτηριστικά μας και την εμπειρία μας. Ας περάσω λοιπόν στα τρία σημεία που είχα προεξαγγείλει. Ε, ο αντίκτυπος παρά τις ε, δυσκολίες η πολιτική συνοχή είχε και σε μακροοικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ορατών αποτελεσμάτων θετικό αντικτύπο για την τσεχική δημοκρατία. Έχουμε μελέτες και από ανεξάρτητους οικονομολόγους που δείχνουν ότι η πολιτική συνοχή είχε πολλαπλαστική ουσιαστικό ε, δίκτυο 0,3%. Δηλαδή κάθε ευρώ της πολιτικής συνοχής προσφέρει 1,3 ευρώ ε, ανάπτυξη στην, ε, ή αποτέλεσμα στην οικονομία της Τσεχίας. Και αυτό είναι και λογικό γιατί η οικονομία μας αντιστοιχεί στο 0,3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ αλλά οι επιχειρήσεις μας εξαρτώνται, οι περιοχές μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δημόσιες επενδύσεις ποσοστό το οποίο σε άλλες χώρες, Πολωνία, Ουγγαρία ή Πορτογαλία είναι πολύ πιο χαμηλό. Έτσι λοιπόν η μία απορρόφηση, η μη απορροφηση η μη απορρόφηση κονδυλίων θα μπορούσε να υπονομεύσει και την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα κονδύλια που δαπανήθηκαν, που απορροφήθηκαν και θα αναφερθώ εδώ και στην μελέτη την πολωνική για το οικονομικό όφελος, για κάθε ευρώ λοιπόν της πολιτικής συνοχής τα 65 λεπτά επανέρχονται σε ευρωπαϊκά κράτη των 15, δηλαδή την Αυστρία, Γερμανία, Γερμανία κυρίως, που ε, ωφελούνται περισσότερο από την αύξηση των εξαγωγών τους προς την Τσεχία. Δηλαδή δεν αποβαίνουν μόνο ο όφελος της χώρας στην οποία επενδύονται άμεσα. Συγκεκριμένα και ορατά απτά αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει χάρη στην πολιτική συνοχή από το 2004. Πάνω από 1.000 θέσεις έχουν δημιουργηθεί. Πάνω από 100.000 θέσεις έχουν δημιουργηθεί χάρη σε αυτά τα προγράμματα. Έχουμε σημαντικές ε, σημαντικά επιτεύγματα με 200 νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις, πολλά κέντρα έρευνας και τεχνολογίας και ανάπτυξης, ε, τα οποία αξιοποιούν και πανεπιστήμια και άλλα ε, άλλοι φορείς. Γενικά δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη διάχυση του αποτελέσματος. Εάν επισκεφθείτε την τσεχική δημοκρατία θα δείτε ότι οι μεταφορές έχουν ιδιαίτερα ωφεληθεί για να διευκολύνονται οι μεταφορές εμπορευμάτων από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία ε, έχουν εξασφαλιστεί απαραίτητες υποδομές και έχουμε μειώσει σημαντικά το διοικητικό φόρτο στην καθημερινή ζωή του πολίτη, στο και αν αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο ορατό. Έχουμε μια σειρά από σημεία επαφής του πολίτη με την διοίκηση, κέντρα εξυπηρέτηση, τα οποία σημαίνουν ότι δεν είναι υποχρεωμένο ο πολίτη να μεταβαίνει είτε στην πρωτεύουσα είτε στι μεγαλύτερε πόλει. Μπορεί να πάει είτε στο εγκύτερο ε, ταχυδρομικό κατάστημα είτε σε οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο εξυπηρέτηση για να ε, ολοκληρώσει διοικητικέ ε, διατυπώσεις που έχει. Ένα άλλο και γενικότερο ζήτημα είναι αυτό της ανάπτυξης των θεσμικών ε, νοοτροπιών και δυνατοτήτων. Αξιοποιούμε την στρατηγική, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση και σε άλλους τομείς, όχι μόνο δηλαδή την πολιτική συνοχής. Και οι φορεί μας γίνονται πιο αποτελεσματικοί γιατί βελτιώνει την ποιότητα της υπηρεσία που προσφέρει ε, η διοίκηση. Υπάρχουν προδιαγραφέ ορισμένες που πρέπει να, να, επι... να επιτυγχάνονται ε, διαφορετικά ε, υπάρχουν συνέπειες. Και βέβαια έχουμε μια θετική και ε, ίσως όχι τόσο από τη συνέπεια που είναι η γενική βελτίωση της διοίκησης, αλλά αυτό είναι κάτι που θα είναι ορατό ε, σύν χρόνο. Αξιοποιούμε λοιπόν τα διδάγματα από τις ε, βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών, κρατών τα οποία Οφελούνται από την πολιτική της συνοχής ή κρατών που ε, έχουν μεγαλύτερη ιστορία. Πάντως είναι κάποια αποτελέσματα λιγότερο απτά και ίσως περισσότερο μακροπρόθεσμα. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν της παρατήρησης ήταν αυτή, αυτό. Ε, τώρα για την πρακτική υλοποίηση, πέρα από τα 2.000 έργα τα οποία με, με το θετικό αντίκτυπο ε, έχουν προχωρήσει ολοκλήρωση. Έχουμε και προβλήματα και δυσκολίες με ενδογενή χαρακτηριστικά την απουσία της ε, παράδοσης ε, της διοικητικής, του, της οργάνωσης διοικητικής, την αστάθεια του διοικητικού μηχανισμού, λογιστικά προβλήματα και εσφάλματα με συνέπειες ε, κυρώσεις, οποίες χρειάστηκε να, ε, να υπομισθούμε, με ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετρήσεις και μέτρα που ε, λαμβάνονται για να επιταχυνθεί η, απο, η λειτουργία της διοίκησης, η βελτίωση του συστήματος για τις δημόσιες ε, προμήθειες και διαγωνισμούς, και το σύστημα προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται με το κόστος του βέβαια αλλά και με τις καθυστερήσεις του. Σημαντικό για μας, πάνω απ' όλα είναι να δεσκόμαστε από τα σφάλματα και να προχωρούμε προς τα βρός. Δεν θα, υπε... δεν θα παραλάβω αυτό είπε ο Πολωνός συνάδελφος. Με μεγάλη εντατικότητα προετοιμάζουμε την προσεχή προγραμματική περίοδο με μια νέα στρατηγική, νέες αρχές. Θέλουμε να επικεντρωνόμαστε σε πιο στρατηγικούς στόχους, εξετάζουμε την, τη λογική της παρέμβασης, θέλουμε να αποφύγουμε την στρεβλωτική ενδεχομένω λειτουργία των ε, πόρων αυτών για την αγορά. Έχουμε μια ενιαία μεθοδολογία που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση με τίτλο περιβάλλον, επικοινωνία με τους ε, δικαιούχους ε, της υποστήριξη κατά τρόπο μηχανογραφημένο πλέον, ηλεκτρονικό μπορούμε να, να εξασφαλίσουμε καλύτερη λειτουργία των, ε, ταμείων, των κονδυλίων της συνοχής που θα λαμβάνουμε και στο μέλλον και πιστεύω ότι έχουμε βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό το δυναμικό και την αποτελεσματικότητά μας. Και τώρα περνάω στο τρίτο σημείο της ε, παρουσίασής μου, όπως ανέφερα στην αρχή. Έχουμε δηλαδή πέραν των εσωτερικών ε, ενδογενών παραγόντων και κάποιους εξωτερικούς που μπορεί να εμποδίζουν την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής όπως θα τη θέλαμε. Έχουμε πέντε χρόνια τώρα οικονομική κρίση η οποία έχει πλήξει σημαντικά την ε, τσεχική οικονομία. Είμαστε ανοιχτή οικονομία όπως σας είπα, είμαστε χώρα διαμετακόμισης και τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώνεται η ύφεση και ε, μακροοικονομική τίτλη αρνητική πλημμύρες επίσης και μέσα στο καλοκαίρι μια άλλη φυσική καταστροφή η οποία σήμανε και ε, έφερε μάλλον και καθυστερήσεις ως προς την, ε, τις υποδομές που προσπαθούμε να κατασκευάσουμε αλλά και επιπλέον επιβάρυνση ως προς την κρατική διοίκηση. Και κάτι ακόμη, και νομίζω ότι σε αυτό είναι πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λόγω των επικρίσεων του ε, ελεγκτικού συνεδρίου, προσπαθούμε να βρούμε μία μέση οδό και να δίνουμε λύσεις ε, οι οποίες μπορεί να μην είναι και να αποφεύγουμε μάλλον ε, τις προτάσεις οι οποίες δεν είναι εμπεριστατωμένες ε, ή επακριβείς. Αυτό το λέω γιατί βλέπω το εκρεμές να μας οδηγεί σιγά σιγά στο μηδενικό σφάλμα. Αλλά αυτό ε, δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα της διόρθωσης και των προσπαθειών μας τόσο, όσο περισσότερο το ότι κανείς θα τολμάει πια να ε, ασχοληθεί με την πολιτική της συνοχής. Έτσι λοιπόν πρέπει να καλύψουμε τους φορείς μας, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στήριξη και προστασία στους φορείς που έχουν διαχειριστεί κονδύλια και μετά την περίοδο των ε, ελέγχων. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα προτιμούσαμε να μην υπάρχει αναδρομική κύρωση, αλλά ε, ε, έγκαιρος έλεγχος της διαχείρισης των κονδυλίων. Αυτό το λέω γιατί σε μια αναφορά στην έκθεση των ε, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου αναφέρεται ότι χρειάζεται βελτίωση της εκτέλεσης. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει αυτές ε, οι ε, πολιτικές να κρίνονται ως προς την ποιότητά τους μόνο από την ανάκτηση κονδυλίων. Και αυτό το, φέρνω σαν πληροφορία και σαν ανατροφοδότηση και από το, το πεδίο αυτό της εφαρμογής των ταμείων συνοχής. Το να δείξουμε πιο αυστηρή στάση απέναντι στη διαχείριση των κονδυλίων δεν θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και την παραγωγικότητα. Για να ολοκληρώσω λοιπόν και για τις κατευθύνσεις που θα παρευτεί η πολιτική στο μέλλον, θα πρέπει καταρχάς να ε, προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την υλοποίηση της πολιτικής, αυτό είναι το σημείο κλειδί, αλλά βέβαια να μην ε, είναι και άχρηστη η υπερητά ε, τα αντικείμενα αυτής της πολιτικής πρέπει να έχουν ουσία και αξία. Και επίσης θα πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο αυτήν την πολιτική, γιατί είναι το μόνο ορατό για τον πολίτη ε, έργο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νέες προτάσεις που κρίνουν πολύ ε, λογικές και εύστοχες. Ε, πρέπει επίση να αποφύγουμε να αποστείλουμε σφαλμένα μηνύματα, αρνητικά μηνύματα δηλαδή, και αυτό το λέω και ενώπιση των ευρωεκλογών. Πέραν των δομικών, διαρθρωτικών μάλλον προβλημάτων, έχουμε μια κυκλικότητα σε αυτή την κρίση και νομίζω ότι η πολιτική της συνοχής είναι ένα κρίσιμο εργαλείο, ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να στηρίξει τις δημόσιες ε, επενδύσεις, μπορεί να βοηθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασία, να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, να δώσει όθηση σε μια ανάκαμψη συστημικού χαρακτήρα. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να κάνω μια στιγμή παρατήρηση, μου επιτρέπετε. Και τη σημερινή ψηφοφορία δεν άνοιξε το δρόμο για μια ευρύτερη ψηφοφορία. Θέλω να ευχαριστώ τον, κύριο Βλασάκ και την Επιτροπή σας για την ε, στάση του στο θέμα αυτό. Αν και πρέπει να σημειώσω ότι μας απογοητεύει το τελικό ε, αποτέλεσμα, η έκβαση τελικά του θέματος, διότι λυπούμαστε που δεν ζητούνται επιπλέον διευθυντικές αλλαγές πρόσθετα κονδύλια. στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά και σε άλλε προτάσεις. Τα συμπέρασματα του Συμβουλίου είχαν πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα με επίδραση και στο πολιτισμό νομικό πλαίσιο. Φαίνεται το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας να έχει απλώς ακολουθήσει άκρητα ορισμένες ε, ε τοποθετήσεις εγώ θα θέλω να επισημάνω ότι πρόκειται εδώ για το σημείο πάνω στο οποίο θα κριθεί η πολιτική συνοχής. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να αποστείλουμε θετικά μηνύματα προς τους πολίτες για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και το θετικό τους αντίκτυπο. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να μεγενθύνουμε, να διωγγώσουμε τον αντίκτυπό τους. Όπως είπε και ο να συνάδελφος, προσπαθούμε να κλείσουμε το χειρότερο δυνατό τις διαπραγματεύσει. και αν είναι να αφαιρθούν μακροοικονομικές αιρέσεις, τότε θα πρέπει κάθε όποια λύση προταθεί να παρακολουθείτε από πολύ μεγάλη προσοχή. Τελικό μου μήνυμα όμως, ας, ε, θα, θα έλεγα στο τελευταίο μήνυμα, ας κλείσουν το ταχύτερο δυνατό οι τριμερείς διάλογοι. Για το χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να αποστείλουμε στον Ευρωπαίο Ψηφοφόρο είναι ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εκκίνηση νέων προγραμμάτων ε, μέσα στα χρονικά πλαίσια, δηλαδή το 2014. Αυτό θα είναι το χειρότερο μήνυμα που θα, μπορούσαν, ε, θα μπορούσαμε να αποστείλουμε. Η πολιτική της συνοχής λοιπόν έχει, για να ολοκληρώνω, ορατά αποτελέσματα, έχει σημαντική προσθεμένη αξία, υπάρχουν ε, περιπλοκές και δυσκολίες προς την υλοποίηση, ιδιαίτερα στην τσεχική δημοκρατία όπου, τα οποία μας προσπαθούμε και να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα με υψηλό κόστος. Είμαστε ωστόσο αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε μια πιο αποτελεσματική πολιτική και να συμβάλλουμε στην Ευρώπη του 2020. Είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε σταθερότητα των κανόνων. Θέλουμε την, η κοινή λογική να επικρατεί σε σχέση με την αντιμετώπιση του δικαιούχου. Θέλουμε μια εξισορρόπηση μεταξύ του αυστηρού ελέγχου και της καταπολέμησης των σφαλμάτων. Αλλά νομίζω και αυτό είναι και ο κρίσιμος ρόλος της Επιτροπής, της Επιτροπής σας, θα πρέπει αυτά να συζητούνται σε εταιρική σχέση με την Επιτροπή, με την Κομισιόν. Και εν τέλει θα ήθελα να υπογραμμίσω το στόχο αυτής της πολιτικής, να βοηθά δηλαδή τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη της συνεργασίας και την ανάπτυξη, την οικονομική. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι το μέλημά μα και ελπίζω να μα βοηθήσετε και εμεί να μπορούμε να σα βοηθήσουμε από πλευρά μα στην υλοποίηση αυτού του στόχου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, λέει ο Πρόεδρο. Καταρχά, ο Γιάννη Όλμπρεχτ έχει το λόγο. Ναι, σα ευχαριστώ και του δύο μιλητέ γιατί είναι θετικό το σημάδι ότι μετά τη γενική δήλωση για το πόσο καλή είναι η πολιτική συνοχή, πλέον έχουμε και κάποια πιο συγκεκριμένα μηνύματα από πλευρά σα και ασφαλώ ε, αυτό μπορεί να είναι προ ικανοποίηση και όχι κάποιων συναδέλφων. Νομίζω όμω ότι για να περάσουμε στο ψητό. Κύριε Υπουργέ, εξηγήσατε τα προβλήματα. Να σας ρωτήσω το επίπεδο των σφαλμάτων μεταξύ της χώρας σας ή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι τυχαίο ή αποτελεί πολιτική στρατηγική. Ήμουνα και στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Δεν είναι το θέμα αν είναι καινούριο ή παλιό το κράτο μέλος. Θα μιλήσω πολωνικά. E, Η πολωνική θέση για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα προκαλεί μεγάλες αμφισβητήσεις και διχογνωμίες εδώ στην Επιτροπή και αυτή η επιχειρηματολογία της πολωνικής ε, κυβέρνησης την οποία παρουσιάσατε, εκεί μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τιμωρούμαστε εμείς. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, γιατί όλα αυτά προέρχονται και από το Μάστρεχτο, όπου εκεί ορίστηκαν οι μακροοικονομικές κυρεώσεις σε ό,τι αφορά και, τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα και τα πράγματα λειτουργήσαν ξεκάθαρα. Επιπρόσθετες λοιπόν επιβαρύνσεις μέσω των κυρώσεων αυτών μπορούν όλα αυτά να υπονομεύσουν την πολιτική συνοχή. Συνολικά θα έλεγα ότι ως Πόλωνος δεν προσυπογράφω όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να τιμωρηθούμε μόνο εμείς αλλά και άλλοι. Αυτό δεν ακούγεται πολύ καλά. Να τιμωρηθούν δηλαδή και άλλοι. Όχι. Θα πρέπει να πετύχουμε μια λογική συμφωνία, μια λογική λύση και φυσικά πάνω απ' όλα να λάβουμε υπόψη τα θέματα αποδοτικότητας. Θα ήθελα λοιπόν ε, να πω ξεκάθαρα ότι η επιχειρηματολογία αυτή της ε, πολωνικής κυβέρνησης, όχι μόνο εμείς αλλά και οι άλλοι να τιμωρηθούν, δεν είναι πολύ πιστική. Να κάνω λοιπόν μια ερώτηση προς τον Υπουργό στην Τσεχία, στην Πολωνία. Έχουν ε, εισαγάγει οι περιφέρειες αντίστοιχες δομές. Το 2013 μέχρι το 2020. Στην περίοδο αυτή πώς ε, θα ορίσετε τα θέματα σωματείων και ευθυνών του, Η επόμενη ομιλητρία, η κυρία Κολάρσκα Κολάρσκα-Ποβίνσκα. Να ευχαριστήσω τους υπουργού που ήρθαν εδώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά ερωτήματα. Ε, σε λίγο θα κλείσουμε την, τα 10 χρόνια από τότε που μπήκαν οι χώρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το εξετάζουμε και από αυτή την οπτική γωνία. Θεωρείτε ότι ένα από τα αίτια μάλλον ένας από τους στόχους της πολιτικής συνοχής έχει επιτευχθεί ο ρόλος δηλαδή των ταμείων σε ό,τι αφορά τη μείωση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών, όχι χωρών μεταξύ περιφερειών, γιατί μιλήσατε και είπατε ότι ένα ευρώ αυξάνει την παραγωγή της οικονομίας, την απόδοση της οικονομίας. Τι γίνεται όμως μεταξύ των φτωχών και πλούσιων περιφερειών μέσα σε ένα κράτος μέλος. Ευχαριστώ, κυρία Σμόλκοβα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω να κάνω και να απευθύνω και στους δύο. Καταρχάς, να ξεκινήσω και να θέσω την εξή ερώτηση προς τον κύριο Μπράουν. Κλείνοντας ε, την παρουσίασή του ανέφερε την πρωινή μας ψηφοφορία. Να τον ρωτήσω αν είναι καινούριο στην κυβέρνηση ή αν συμμετείχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Νέτσας. Γιατί αν συμμετείχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει ενημερώσει το ότι στην συνεδρίαση του Φεβρουαρίου θα μπορούσε να έχει ζητήσει κάτι άλλο πέρα από τα 900 εκατομμύρια στο νησιν Μία άλλη ερώτηση όμως. Είναι γνωστό ότι η Τσεχία και η Πολωνία είναι κράτη-μέλη όπου η κατανομή των ε, πόρων και των ταμείων δεν αποφασίζεται μόνο από την κυβέρνηση και από τα μεμονωμένα υπουργεία, όχι δηλαδή μόνο σε κεντρικό επίπεδο, αλλά τμήμα των πόρων ε, ανατίθεται και διανέμεται από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Πείτε μας, τι πιστεύετε, τι ποσοστό των πόρων αυτών είναι λογικό και χρειάζεται για την πολιτική συνοχή προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, να είναι άμεση, καλύτερα ελεγχόμενη, με καλύτερα αποτελέσματα και επίσης να αποτρέψει την διαφθορά. Με το αναφέρατε αυτό, αλλά το ξέρουμε από τον τύπο ότι κάποιες χώρες θα πηγαίνουν καλύτερα, κάποιες χειρότερα. Όταν λοιπόν ε, δίνουμε τους πόρους αυτούς και τους δίνουν μάλλον οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, ε, είναι δυνατόν να υπάρχει καλύτερη έτσι χρήση των πόρων. Ευχαριστώ. Βίκτορ Μποστινάρο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους δύο πολύ σημαντικούς ομιλητές. Είχα το προνόμιο να συνεργαστώ στενά με τους εκπροσώπους της πολωνικής κυβέρνησης ως εισηγητής και επίσης έχω συνδεθεί με τον κύριο Μπράουν τουλάχιστον δύο φορές. Ήταν πραγματικά πολύ επιτυχής αυτή η εμπειρία τότε, πολύ καλύτερο και πολύ καλύτερη από κάθε άλλη εμπειρία που είχα με την πρώην ρουμανική κυβέρνηση. Αυτό το λέω και το τονίζω. Δεύτερο σημείο. Να τονίσω το ρόλο που διαδραματίζει σήμερα η Πολωνία για την πολιτική συνοχή. Εν γέννη. Γιατί από το πολύ καινοτομικό σχέδιο μέχρι το αφηρημένο ε, επίπεδο της πολιτικής συνοχής πρόκειται για μία από τις κορυφαίες εμπειρίες που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη. Εγώ Ρουμάνος είμαι, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερος που βλέπω μία χώρα που μπήκε μετά το 2004 στην Ένωση να γίνεται ηγετική, ανταγωνιστική, κινητήριος δύναμη για τη βελτίωση, την καινοτομία της πολιτικής συνοχής. Και αυτό καταδεικνύει ότι ακόμα και τα καινούργια μέλη σε κάποιες περιπτώσεις θα πηγαίνουν και καλύτερα ακόμα από τις παλιές χώρες. Ένα άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω. Θα διαφωνήσω λίγο με αυτό που είπε ο κύριος Μπράουν. ότι ο υπερβολικός και είναι επιβλαβής για την πολιτική συνοχή. Να είμαστε σαφείς το αποτέλεσμα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου, αλλά και αυτός ο υπερβολικός διακυβερνητισμός ήταν βασικός εχθρός της μελλοντική διάστασης της πολιτικής συνοχής. Και αυτό θα το βελτιώσουμε όλοι για το μέλλον. Είναι ένα μάθημα το οποίο ίσως να μην αρέσει σε όλους, αλλά αληθεύει ότι το Κοινοβούλιο έκανε ό,τι μπόρεσε για να ξεπεράσει αυτή την κληρονομιά της διακυβερνητικού χαρακτήρα. Τώρα, μία μικρή ρουμάνικη εμπειρία μετά τη δική σας ε, παρέμβαση που ήταν πολύ σημαντική για όλους μας. Καταρχά, στη Ρουμανία, και αυτά είναι τα πορίσματα μίας μελάτης, την οποία εγώ έδωσα την εντολή να γίνει για τη χώρα μου, σε ό,τι αφορά την νομική και τη θεσμική αβεβαιότητα. Το ανέφερε και ο Τσέχος ομιλητής. Αλλά στην Ρουμανία αυτό είναι πολύ πιο βαθύ ως ε, φαινόμενο και πολύ πιο επιζήμιο για την πολιτική συνοχή. Η πολιτική ανάμειξη και η σχέση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και το, της πολιτικής πελατείας με δραματικό αντίκτυπο και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και ό,τι αφορά τον ρόλο των ελεγκτικού συνεδρίου σε επίπεδο Ρουμανίας αλλά και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η απόφαση να ανασταλούν έξι ε, προγράμματα, επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι 6 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικής αξίας. Δραματικό αυτό για την περίοδο 2009-2011. Δραματικό, δραματικό αυτό το μάθημα που αναγκάστηκε να μάθει η Ρουμανία. Έλλειψη στρατηγικής. Χαίρομαι, χαίρομαι και με εμπνέει πάντα το πολωνικό μοντέλο, ειλικρινά. Είμαι υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της πολιτικής συνοχής. Με εμπνέει λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο η Πολωνία καταρτίζει στρατηγικές για το μέλλον της χώρας. Αλλά στην περίπτωση της Ρουμανίας δεν υπήρξε πραγματική στρατηγική. Μόνο κάποια επίπλαστα στοιχεία. Η συγχρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τώρα την κρίση, όχι μόνο στη Ρουμανία αλλά και σε άλλες χώρες. Δραματικές ήταν οι συνέπειες. Έλλειψη συγχρηματοδότησης και δημοσιονομικού προϋπολογισμού, ε, σχεδιασμού για μία περίοδο ενός έτους σε ό,τι αφορά πολιτικές που παίρνουν πολλά χρόνια. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει πολιετή σχεδιασμό σε ό,τι αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότηση. Το αντιμετωπίζει η Ρουμανία αυτό το πρόβλημα. Κάτι άλλο. Μεγάλε ελλείψει σε ό,τι αφορά το διοικητικό και το θεσμικό επίπεδο. Στην Πολωνία και στην Τσεχία υπάρχουν ε, υπηρεσίε, θεσμικά όργανα που είναι έτοιμα να εφαρμόσουν, να καταρτήσουν, να ελέγξουν την πολιτική αυτή. Στη Ρουμανία να μην προσθέσω και άλλα ονόματα σε αυτόν τον ε, επόδυνο κατάλογο, αλλά είναι και άλλες οι χώρες αυτές. Έλλειψη, έλλειψη απόδοση σε ό,τι αφορά το διοικητικό επίπεδο των υπηρεσιών. Αυτό μεγάλο, μεγάλο πρόσκομα σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή. Εδώ κάπου θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ και πάλι θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή είναι τόσο σημαντική, όχι μόνο για να εξαγάγουμε τα μαθήματα από αυτά που είδαμε στο παρελθόν, αλλά γιατί, όπως είπαν και ο κύριος Μπράουν και ο, ο Υπουργός Μπράουν και ο κύριος ε, από την πολιτική κυβέρνηση, αυτά θα τα πετύχουμε μόνο βάσει των ίδιων κριτηρίων και προτύπων με ίδια μέτρα και σταθμά και να μην υπάρχουν τέτοιες ε, διακρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η πρόεδρο. Τώρα έχουμε τρεις ομιλητές, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι και να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και εδώ κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Χόιμπνερ, να ευχαριστήσω τους Υπουργούς ε, της Πολωνίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και θα ήθελα στη συγκεκριμένη περίπτωση να αναφερθώ στην πολύ χρήσιμη διαδικασία και που είχε η Κροατία και με τις δύο κυβερνήσεις και επίσης να σας πω ποιες ήταν οι εμπειρίες που είχαμε μεταξύ της, Κροατίας και της Πολωνίας. Πολύ χρήσιμη συνεργασία. Υπογράψαμε μία, συναντήση, μία συμφωνία μεταξύ τεσσάρων ε, επαρχιών της Κροατίας και αντίστοιχων ε, πολωνικών. Όλες αυτές οι εμπειρίες λοιπόν στην Πολωνία έχουν ενδυναμώσει την ικανότητα της Πολωνίας να αφομοιώσει τους πόρους των ταμείων συνοχής. Όλα αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε στα επόμενα χρόνια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο παρά το γεγονός ότι το μέγεθος της χώρας διαφέρει τόσο πολύ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν ισχύουν απαραίτητα οι ίδιες συνταγές που χρησιμοποιήσατε εσείς και στη δική μας περίπτωση. Αλλά επειδή επειδή θα έχουμε πάνω από 1,2-1,3 δισεκατομμύρια την επόμενη πολιετή περίοδο, θεωρούμε ότι για να υπάρξει μεγαλύτερη απορρόφηση και ανάπτυξη των Ταμείων συνοχή, καλή θα είναι η ανταλλαγή τέτοιων εμπειριών με την Κροατία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο κυβερνήσει για την έω τώρα συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλάσακ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω πόσο εκτιμώ τις παρουσιάσεις αυτές των υφυπουργών και να αναφέρω ένα σημαντικό στοιχείο. Πολλά μάθαμε από την προηγούμενη περίοδο. Νομίζω ότι η προσέγγιση της κυβέρνησής μας ε, για την επόμενη περίοδο είναι καλύτερη. Μείωση του αριθμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων από 24 σε 8 στον αριθμό. Μία ενιαία μεθοδολογία για κάθε πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα ενημέρωσης σε κάθε χώρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την μελλοντική περίοδο. Ρωτώ λοιπόν, αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν συζητάτε θέματα νομοθεσίας. Θεωρείτε ότι υπάρχουν προκλήσεις, απειλέ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Τελευταίο ο Η ομιλήτρια μάλλον. Η κυρία Μαλετίτς θα σας ευχαριστούσα κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους εκπροσώπους της κυβέρνηση της Τσεχίας και της Πολωνία. Έχω κάποιε ερωτήσει να σα κάνω. Καταρχάς, ό,τι αφορά τα μέτρα σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τέτοιων σχεδίων, σε ό,τι αφορά την προχρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση. Πώς διαμορφώθηκαν τα α, χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποίησατε. Πώς ε, συνδυάζετε τα μέτρα ε, λιτότητας και τα μέτρα δημοσιονομικών περικοπών με τα μέτρα εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, αυτές οι εμπειρίες για μας στην Κροατία. Πείτε μας κάτι παραπάνω. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των σχεδίων. Έχετε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία των προγραμμάτων για το 2020. Ξέρετε ότι ακόμα προετοιμάζετε επιχειρησιακά προγράμματα και άλλα στρατηγικά έγγραφα, αλλά κάποια κεφαλαϊκά προγράμματα χρειάζεται να προετοιμαστούν πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν θα με ενδιαφέρει να μου πείτε πότε, αν έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία. Ο κύριο Γκουτμάνης και κλείνουμε το... Έχει κλείσει ο κατάλογος. Να είστε πολύ σύντομο, Όχι, όχι, παρακολούθησα τις δύο παρεμβάσει, πάρα πολύ προσεκτικά. Ναι, ναι, λέει η πρόεδρο. Μία ερώτηση προ τον Τσέχο Υπουργό. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει στα αλήθεια οι πληρωμές ακόμα και για τα κοινωνικά ταμεία που δεν αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό του συνόλου σταματούν. Σταμάτησαν. Το 2011 δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και σταμάτησαν και το 2012. Και ακόμα και τώρα, κοιτώντα τι γίνεται, στη τσεχική δημοκρατία είδω ποσοστό απορρόφησης χωρίς καμία διαφορά από το Φεβρουάριο, στον τελευταίο χρόνο. Ποτέ δεν αυξάνεται η απορρόφηση από 1η Ιανουαρίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ίδιο αναπεριοχή. Η τελευταία χρονική στιγμή τον Ιούλιο ξαφνικά βελτιώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες η απορρόφηση. Είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε αυτά, γιατί η έκθεση του ιριού Βλάσακ που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα που υπάρχει με τη δέσμευση θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ σημαντικό για χώρες ε, σημαντικές και για άλλες ε, και οι Τσέχοι και η Ρουμάνοι αν δεν επιτραπεί δηλαδή μεταφορά το 2011, 2012 και 2013. Είναι εσωτερικέ αυτέ οι πληροφορίε. Αλλά πείτε μου, από πλευρά μεθοδολογία, τι λόγοι υπάρχουν. Πολιτική μεθοδολογία, η Πράγα λαμβάνει επιπλέον πόρου. Ωστόσο, το σύνολο τη τσεχική δημοκρατία θα χάσει. Το επόμενο φάκελο είναι 22% μικρότερο από ό,τι ω τώρα. Τι λόγος υπάρχει λοιπόν γι' αυτό, γιατί από άλλες πτυχές είσαστε μία από τις καλύτερες χώρες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, να δώσω το λόγο στους υπουργού να πάρουν το λόγο όπως τον επιθυμούν για να απαντήσουν τις ερωτήσεις. Η Δημοκρατία, κύριε Τάνιλ Μπράουν, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε και για το feedback, αν και Κάποια σχόλια ήταν αρκετά σκληρά. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος καθότι από ό,τι καταλαβαίνω ε, έχουμε πίεση χρόνου σε ό,τι αφορά τα δύο πρώτα θέματα τα οποία αλληλοσυνδέονται για το ρόλο των περιφερειών. Τι ποσοστό θα πρέπει να αφιερωθεί και να δοθεί στο περιφερειακό επίπεδο και ποιος είναι ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Ταμείων σε ό,τι αφορά και τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών και ποιος είναι ο ρόλος των ε, περιφερειών στη διαχείριση των πόρων. Καταρχάς, οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών έχουν και μειωθεί και αυξηθεί. Νομίζω ότι ο εμπειρογνώμονος θα μπορούσε να σας το εξηγήσει αυτό, αλλά γενικά σε επίπεδο περιφερειών, ΝΑΤΣ 2, οι διαφορές έχουν μειωθεί. Αυτό συνάδει, θεωρώ, με τη γενικότερη τάση που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών. Οι διαφορές μειώνονται, αλλά σε υποπεριφερειακό επίπεδο οι διαφορές από την άλλη έχουν αυξηθεί τα τελευταία 10 χρόνια στη ζωική Δημοκρατία, έγινε αυτό και γι' αυτό δεν εξετάζουμε καταρχάς το ρόλο των Δήμων και των κοινοτήτων σε ό,τι αφορά την διαχείριση, αλλά προσπαθούμε να επικεντρώσουμε τις επενδύσεις σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Κοιτάμε λοιπόν ενοποιημένες προσεγγίσεις, κοιτάμε τις περιφερειακές διαφορές. Δεν είναι βασικά θέμα διαχείρισης, είναι θέμα πολυεπίπεδη και κυβέρνηση. Και για μα η περιφερειακή πτυχή διάσταση τι σημαίνει ότι γίνεται διαφοροποίηση σε υποπεριφερειακό επίπεδο και σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων. Η απόφαση λοιπόν της κυβέρνηση ήταν η εξή Μείωση του αριθμού των προγραμμάτων για πολλούς λόγους, διοικητικού λόγω θεσμικών ε, ρυθμίσεων, αλλά εξετάζουμε στενά τα θέματα τα οποία θα συμμετέχουν στο επόμενο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Τώρα έχουμε περίπου 18% ε, έχουμε προγράμματα τα οποία έχουν ε, το 18% των πόρων και έχουμε και θεματικά ζητήματα, θεματικά ναι. προγράμματα. Έξι θεματικά προγράμματα σε κάθε εξ αυτών εξετάζουμε τους συγκεκριμένους όρους, προσπαθούμε να πετύχουμε μια συμφωνία με τους περιφερειακούς εταίρους και αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Τι σημαίνει η περιφερειακή ανάπτυξη, τι σημαίνει μια ανοποιημένη προσέγγιση. Σημαίνει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο περιφερειών. Ποιο είναι το εργαλείο, μια ανοποιημένη προσέγγιση ή μια πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Αυτό είναι που μας απασχολεί. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να χάσουμε τις διοικητικές ε, ικανότητες στην περιφέρεια. Αυτές θα παραμείνουν. Τα ποσοστά και η δομή είναι ακόμα υποσυζήτηση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η περιφερειακή διάσταση θα είναι κατά ποσοστό λίγο μεγαλύτερη από ό,τι στην τρέχουσα περίοδο, 25-30%. Είναι υποσυζήτηση όμως αυτό και οι συζητήσεις υπησέρχονται σε λεπτομέρειες με τους υπουργούς για να προσπαθήσουμε να δούμε ποιος είναι ο στόχος στο περιβάλλον, για παράδειγμα, μείωση των ε, εκλειόμενων αερίων, από πού προέρχονται τα αέρια αυτά, τι χρειάζεται σε κάποιες περιπτώσεις, ε, διαφοροποίηση και το καθεξής. Και σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και αποφάσεις, λαμβάνονται αποφάσεις για την ε, θεσμική λειτουργία των υπηρεσιών. Για την ερώτηση της κυρίας Κολάρσκα τώρα για το κατά πόσο ο ρόλος των ταμείων ε, των ευρωπαϊκών μπορεί να έχει να κάνει και να πετύχει την μείωση των διαφορών. Νομίζω ότι υπάρχει μια τάση να εστιαζόμαστε πιο πολύ στην ανάπτυξη και στην απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η πολιτική συνοχή να αποτελεί ένα εργαλείο για την επίτευξη των στόχων τη Ευρώπη του 2020 σε ό,τι αφορά και τέτοια ζητήματα συνοχή. Θεωρούμε ότι ο στόχο τη συνοχή θα πρέπει να υπάρχει. Άρα μία από τι πέντε προτεραιότητε για την επόμενη προγραμματική περίοδο μειώσαμε τον αριθμό των ε, προτεραιοτήτων, αλλά ένας από τους στόχους είναι μια ισορροπημένη ανάπτυξη των περιφερειών. Αυτό θα το πετύχουμε αναπτύσσοντας το δυναμικό όλων των περιφερειών αυτών που έχουν διαφορετικές ανάγκες και αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εξισωθεί η απόδοσή τους προς τα πάνω προς τα κάτω. Αναφερθήκατε επίσης σε θέματα διαφθοράς. Δεν το αναφέραμε εμείς, θα το αναφέρουμε τώρα να σας πω ότι το 90% των σφαλμάτων είναι μη θελημένα. Αλλά πρόκειται για μια πλευρά της πολιτικής συνοχής που είναι επιζήμια και για, το, για την εικόνα της πολιτικής και σε εθνικό επίπεδο. Δεν θέλουμε μόνο σε αυτό να επικεντρωθούμε. Κοιτάμε θέματα απλοποίησης, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται και προλαμβάνονται τα μη θελημένα σφάλματα αλλά υπάρχει και η στρατηγική κατά της ε, διαφθοράς που θα εφαρμοστεί στην ε, μεθοδολογία. Χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε και την εμπειρία που μπορεί να μας δώσει η διεθνής διαφάνεια και άλλοι τέτοιοι θεσμικοί οργανισμοί. Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία και την επιλογή των ε, προγραμμάτων, πρόκειται μια πάρα πολύ για μια πολύ επικίνδυνη φάση σε ό,τι αφορά θέματα διαφθοράς και γι' αυτά λοιπόν θα τους δώσουμε τη σημασία τους για την ερώτηση του κ. Βλάσακ για το κατά πόσον ε, θέλουμε να υπάρχει μία ενιαία μεθοδολογία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Πρόκειται για ένα εθνικό εγχείρημα. Και μόνο η εθνική, το εθνικό επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί ε, υπεύθυνο. Δεν νομίζω ότι αυτό υπονομεύεται από οποιαδήποτε διαδικασία εδώ σε ό,τι αφορά θέματα προχρηματοδότηση και προετοιμασία, Έχουμε κάνει μια σχετική ανάλυση και καθ' όλη τη διάρκεια τη περίοδου πώ μπορούμε να βοηθήσουμε του δικαιούχου προκειμένου να μην προβαίνουν στους δανεισμούς, περιτούς, σε ό,τι αφορά την προχρηματοδότηση, χρηματοδότηση δηλαδή εξάντε. Ενέχει κάποιου κινδύνου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του κανόνε περί του προπολογισμού σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, με κυβερνητικέ οργανώσει. Σε κάποιε περιπτώσει χρησιμοποιείται προχρηματοδότηση. Για τι πιο πολλέ περιπτώσει χρησιμοποιείται ένα τροποποιημένο σύστημα πληρωμών, όπου ουσιαστικά οι υπηρεσίε μπορούν να πληρώσουν για τον δικαιούχο μετά από έναν πρώτο έλεγχο. Μπορώ να σα δώσω πιο πολλέ πληροφορίε, αν θέλετε, λεπτομερίε για κάποιε online ε, πληρωμέ. Ναι, τώρα σε ό,τι αφορά τα μέτρα λιτότητα, τα μέτρα περικοπών του προπολογισμού. Είχαμε τέτοια μέτρα. Αλλά μέχρι τώρα, μέχρι τώρα δεν είχαμε σημαντικές ιδέες συγχρηματοδότησης για την Ευρώπη που να μην χρηματοδοτήθηκαν. Ήταν υποχρεωτικό, υποχρεωτική η δαπάνη. Μπορούν λοιπόν να συνάδουν αυτά για την προετοιμασία των project. Να πω δύο πράγματα. Σε συστημικό επίπεδο κάνουμε αξιολογήσεις εξάντια για τα μελλοντικά προγράμματα και τμήμα των ε, αναλύσεων αυτών εξάντε έχει να κάνει με την ανάλυση της ικανότητας απορρόφησης σε ό,τι αφορά την αρχή των project επίσης, τεχνική αρρωγή για τους μελλοντικού ε, κατόχους των κοινωνιοποιημένων προσεγγίσεων. Τέτοιες ε, προετοιμαστικές, προπαρασκευαστικές δράσεις. Για την τελευταία ερώτηση που ήταν πολύ θεωρητική. Ναι, υπάρχει ένας κίνδυνος ε, αποδέσμευσης, αν και αναζητούμε εδώ και καιρό μια συστημική λύση, την οποία όπως ανέφερα εγώ ίδιος, δεν θεωρώ ότι αποτελεί έξυπνη λύση. Η λύση είναι η ε, για τα έτη 2007-2013. Και τώρα για την επόμενη περίοδο και πάλι βλέπω αυτό το 1 3. Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό, τι να πω. Τώρα, το τρέχον έτος έχει μεγάλο κίνδυνο, κίνδυνο ήταν εξ αρχή το 2013 πολύ επικίνδυνο για τις χώρες ε, του Ταμείου Συνοχής. Το λέγαμε αυτό εξ αρχή. Ήταν ε, ένα ωραίο δώρο. Εμείς το εγκρίναμε. Αλλά δημιουργήσαμε έτσι και μια δύσκολη κατάσταση όπου σήμερα θα πρέπει να ξοδέψουμε διπλές ε, δαπάνες και πολύ απλά ούτε η οικονομία ούτε η κυβέρνηση είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Δεν αποφεύγω τα προβλήματα και το ανέφερα και στην παρέμβασή μου ότι έχουμε λάβει ακόμα και δυνηρά μέτρα. Έχουμε, ή αναγκαστήκαμε να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε κάποιες ε, κάποια ελλείμματα και προβλήματα, αλλά ασφαλώς εδώ και καιρό λέμε ότι αναζητούμε μια συστημική λύση και πολύ απλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αν δεν ε, θα πληθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Τον κύριο Κουμπιάκ παρακαλώ τώρα. Θα συνεχίσω από αυτά που είπε ο προηγούμενος, αν και φοβάμαι ότι δεν έχω μείνει και πολλά για να σας πω. Ας ακολουθήσουμε όμως την σειρά των ερωτήσεων. Αρχίζω λοιπόν με το θέμα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Βεβαίως η θέση μας επ' αυτού δεν είναι να τιμωρήσουμε εξίσου όλα τα κράτη-μέλη ή να τα υποβάλουμε όλα στους ίδιους κανόνες. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να υπάρξει μια σωστή διευθέτηση και κανονισμοί, οι ίδιοι κανόνες βέβαια για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά το πρόβλημα του αυξανόμενου ελλείμματος είναι κάτι κοινό στην εποχή μας και πιέζει και τους καθαρούς πληρωτές και όσους εποφελούνται από δάνεια. Η μακροοικονομική αιρεσιμότητα αφορά και εκείνους που δεν τους υποβάλλουμε σε αυτό το κανόνα καθόλου. Σας είχα πει και πριν ότι χρειάζεται φρόνηση στον καθορισμό της σχέσης μεταξύ οικονομικής διακυβέρνησης και χρήσης των κοινοτικών κονδυλίων. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε ακόμη τον χρυσό κανόνα για να συναντηθούμε στη μέση. Αυτό προσπαθούσα να σας πω από πριν. Επόμενη ερώτηση αφορούσε το κατά πόσον τα ευρωπαϊκά ταμεία χρειάζονται, θα χρειάζονται και στο μέλλον όπως χρειάζονται τώρα. Φυσικά, στην περίπτωση της χώρας μου της Πολωνίας, παρατηρήσαμε μία σύγκληση μεταξύ των αναγκών των περιφερειών και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται. Μιλάω για τη σύγκληση όχι μόνο στη χώρα μου, αλλά βέβαια και στον κοινοτικό μέσο όρο. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα χρειαζόμαστε τα ταμεία αυτά και στο μέλλον, έχουν κονδύλια αυτά. Διότι έχουμε σημειώσει μερικές ανισότητες. Θα θέλουμε λοιπόν να συνεχιστούν γιατί στην Πολωνία για πολλά χρόνια η κυβέρνηση τόνιζε ότι τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής ως προς την προώθηση της ανάπτυξης και το γεφύρωμα των αναπτυξιακών χασμάτων και την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων, αυτά ακόμα υπάρχουν και σε περιφερειακό επίπεδο στην Πολωνία, στα κράτη-μέλη και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ναι, θα χρειαστούν, θα συνεχίσουν να χρειάζονται αυτά τα κονδύλια και στο μέλλον. Όχι μόνο η Πολωνία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επεκτείνεται. Υπάρχουν, υπάρχει ένα νέο κράτος μέλος η Κροατία ας πούμε Αυτά τα κονδύλια λοιπόν, αυτά τα ταμεία δεν είναι μόνο για μας τους Πολωνούς ή για τις χώρες που έχουν ήδη μπει από το 2004 ή το 7, Βουλγαρία και Ρουμανία, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που θα προσέλθουν στο μέλλον. Τρίτο θέμα ήταν η αποκέντρωση και η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα ήθελα να πω ότι στην Πολωνία είμαστε πολύ περήφανοι για την αποκέντρωση γιατί τη μεταρρύθμιση που αφορούσε την αυτοδιαχείριση ή μάλλον την τοπική αυτοδιοίκηση την αρχίσαμε ήδη από το 90 στις πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Πολωνία είχε ήδη γίνει λόγος για τη δημιουργία της αυτοδιοίκησης και η διαδικασία αυτή τελείωσε την 1η Ιανουαρίου του 1999 όταν ολοκληρώθηκε το σύστημα μέσω της δημιουργίας των βοηβοδάτων και των περιφερειών. Όταν επισκέπτομαι χώρες σαν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και ίσως και άλλες, Βλέπω ότι θεωρούν την Πολωνία σαν ρότυπο λόγω του υψηλού ρυθμού απορρόφησης των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και τους λέω πάντοτε εμείς χρησιμοποιήσαμε την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Δεν έχουμε μόνο εθνικού επίπεδου προγράμματα, αλλά κάθε βοηβοδάτο είναι μία αυτοδιοικούμενη αρχή. Και γι' αυτόν τον λόγο η απορρόφηση για την Πολωνία είναι 88%. Αυτό το παράδειγμα μπορεί να ακολουθηθεί και από άλλους νομίζω. Και πετύχαμε σε τέτοιο βαθμό ώστε για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα χορηγήσουμε ακόμη περισσότερες δικαιοδοσίες στις περιφέρειες για να διαχειριστούν μόνες τους τα ταμεία, τα κονδύλια αυτά. Να γίνει δηλαδή περαιτέρω αποκέντρωση και θα ορίσουμε το 60% σε σύγκριση με το τωρινό 37% 60% των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής θα δοθούν στις περιφέρειες. Άλλο θέμα για την διαφουθορά, για το κατά πόσον η αποκέντρωση και η χορήγηση εξουσιών στις περιφέρειες δεν δημιούργησε ακόμη περισσότερους κινδύνους διαφθοράς. Δεν το είδαμε αυτό, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Στην Πολωνία τουλάχιστον έχουμε έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς λαθών και απατών. Άμα θέλετε το λέμε και διαφθορά. Άρα η αποκέντρωση στην Πολωνία λειτουργεί. Και γι' αυτό επισκεπτόμενος άλλες χώρες όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και Πολωνία, με ρωτάνε πάντοτε για την αποκέντρωση στην Πολωνία. Αλλά ακόμη και στο Καζαχστάν αν πάω και μιλήσουμε για την καλύτερη δυνατή χρήση των κονδυλίων, είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι από το πετρέλαιο, πάντοτε με ρωτάνε για την αποκέντρωση, για τη μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης ως υπόδειγμα. Στην περίπτωσή μας λοιπόν μπορώ να πω ότι η εφαρμογή των τριών επιπέδων αποκέντρωσης λειτουργήσε υπέρ της σαφήνειας και της ακαιρεότητας. Και φυσικά τα κονδύλια χρησιμοποιούνται, απορροφούνται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Πάντα βέβαια υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να το ανηθούμε αυτό, συμβαίνει και αυτό, αλλά εξε, όλος εξαιρετικός. Τώρα τα σχόλια που ακούστηκαν από τον Ρουμάνο συναδελφό μας και τον Κροάτι από εδώ και από εκεί. Τι να σας πω. Είναι απλώς σχόλια όσο και αν είναι θετικά. Πολύ κολακευτικά για την Πολωνία και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το Υπουργείο μας συνεργάζεται τόσο στενά με τις χώρες αυτές και έχουμε συνεχείς ανταλλαγής επισκέψεων και απόψεων. στέλνουμε εμπειρογνώμονες για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να αποκεντρώσουμε και να απορροφήσουμε περισσότερο τα κονδύλια. Το δέχομαι λοιπόν, ναι, έχουμε τέτοια συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ, Μπάρτζο Τζινκούε. Τα άλλα θέματα νομίζω τα εξάντλησε ο Τσέχος συνάδελφός μου του οποίου συμμερίζομαι την άποψη σε πολλά θέματα και γι' αυτό ας μην συνεχίσω εγώ. Βέβαια, προετοιμάζουμε και καινούργια προγράμματα για την προοπτική μέχρι το 20, 14-20 για στις μεταφορές ας πούμε. Αρχίζουμε διαγωνισμό για την ανάληψη του έργου. Τι άλλο έχω εδώ προχρηματοδότηση, όχι αυτά, αυτά. Αν ξέχασα τίποτε πέστε μου. Ο κύριος Sorry, but I really want to... Γκουτμάνησε. Θέλω να ρωτήσω κάτι και τους δύο υπουργούς για την μακροοικονομική αιρεσιμότητα που θα είναι η τελευταία μάχη που θα δώσουμε στον τριμερή διάλογο σήμερα. Ε, ελπίζουμε να είναι η τελευταία. Εσείς είστε μέλη κυβερνήσεων και οι πρωθυπουργοί σας, τουλάχιστον οι περισβευτές σας, έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση της έννοιας αυτής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Το τελευταίο κείμενο του Συμβουλίου εγκρίθηκε δεν ξέρω με τι πλειοψηφία, και λέει ότι θα χρησιμοποιηθούν δύο και μόνο αρχές για τις μη πληρωμές. Δηλαδή πρώτον αν η χώρα δεν σέβεται τους κανόνες για τα υπερβολικά ελλείμματα η πρώτη προειδοποίηση μείον 50% η δεύτερη μείον 100%. Δεύτερο κριτήριο αν υπάρχουν ανισορροπίες δηλαδή μεγάλο έλλειμμα κλπ επίσης εμπορικό ισοζύγιο. Και εκεί θα κοπούν πολλά χρήματα. Ερωτώ λοιπόν, μα τελικά όλες οι χώρες που συνυπόγραψαν πιστεύουν ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι τόσο ελάχιστα ώστε είναι εύκολη η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων και δεν θα τους εφαρμοστεί και σε εκείνους. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με το Eurostat, το έλλειμμα του 12 ισχύει για 16 χώρες πάνω του 3% και μεταξύ αυτό είναι και η Πολωνία και η Τσεχία. Γιατί λοιπόν τέτοια συνένεση ως προς τα δύο αυτά κριτήρια. Διότι αν η Κομισιόν περικόψει τα ε, μία δεν θα πάρετε τίποτα γιατί για να καλυφθεί το έλλειμμα σημαίνει να κοπούν χρήματα από αλλού, όχι από τα διαρθρωτικά συνήθως ταμεία θα σήμαινε λογικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, πολύ γρήγορα ποιος θέλει να απαντήσει. Η συντομότατη απάντησή μου είναι ότι βέβαια δεν μπορώ να πω ποιος ενέκρινε τα κριτήρια αυτά, αλλά υπάρχουν τώρα, δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε. Δεν θα βοηθούσε αυτό τίποτα να τα ξαναδιαπραγματευτούμε από την αρχή. Αυτό είπα και πριν. Είπατε ότι 16 χώρες έχουν μεγάλο υπερβολικό έλλειμμα. Αυτό προσπαθούσα να πω δηλαδή και εγώ, ότι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο και η επιβολή της μακροοικονομικής ερεσιμότητας μπορεί να μην τους βοηθήσει όλους όσους ωφελούνται από τα κονδύλια. Ίσως ο συνάδελφός μου εδώ έχει να προσθέσει τίποτα. Ναι, δύο σχόλια. Δεν είναι το θέμα που γνωρίζω πολύ καλά βέβαια, αλλά πρώτον, η εφαρμογή των κριτηρίων πρέπει να αποσαφινιστεί τώρα μέσω μιας κατεξουσιοδότησης πράξης όπου θα συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φαντάζομαι θα ξανασυζητηθεί το θέμα. Και έπειτα πιστεύω εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν νομίζω ότι είναι ίση μεταχείριση να συνδέσουμε τα δημοσιονομικά και τα ελλείμματα με μία και μόνη πολιτική, δηλαδή την πολιτική συνοχής. Αυτά ήθελα να σας πω από εθνικής σκοπιάς. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο λίγη η ανταλλαγή απόψεων με τους υπουργούς. Τους ευχαριστώ και τους δύο για την πολύ ενδιαφέρουσα συμβολή τους εδώ στη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ. Επόμενο θέμα το 19. Δημόσια κρόαση για την εμπειρία τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη όσον αφορά την εφαρμογή τη πολιτική για τη συνοχή δύο τελείε διδάγματα που αντιλήθηκαν και μελλοντικέ προοπτικέ τελεία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στον πρώτο εμπειρογνώμονα, τον καθηγητή Τζον Μπάτλερ. Το θέμα του είναι η εμπειρία των κέντρο-ανατολικοευρωπαϊκών χωρών. Έχει το λόγο. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι λόγω του περιορισμού του χρόνου πρέπει να είστε, να είστε σύντομοι και ακριβείς. Αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλησπέρα κυρίες και κύριοι. από το Πανεπιστήμιο Στρόθκλετ της Λασκόβης. Και ήρθα να σας δώσω κάποιες ε, παρατηρήσεις για την εφαρμογή των πολιτικών στην Ανατολική Ευρώπη. Καταρχάς θα υπενθυμίσω σύντομα τι είδους κονδύλια αξιοποιούνται και δεύτερον, Οι 12 χώρες, τις ε, πρώτες 12 χώρες και βέβαια και ευρύτερα στο σύνολό τους ε, η τωρινή Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια για την πολιτική. Χρήσιμο λοιπόν είναι νομίζω το ότι πριν από τη δική μου παρουσίαση ακούσαμε τους δύο υπουργού γιατί έτσι έχουμε μια σαφή εικόνα. της κατάστασης. Οι πιστώσεις που βλέπετε για την πρώτη περίοδο σε πράσινο και για την τρέχουσα σε μπλε έχουν και βλέπετε τη σημασία του για και την Πολωνία ένα συνολικό ποσοστό πολύ υψηλό για τις δύο αυτές χώρες και ως εκ τούτου η επιτυχία της αξιοποίησης των κονδυλίων έχει κεντρική σημασία για όλες τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Δεύτερον, χωρίς να είναι πολύ σαφής η εικόνα όταν δουλεύουμε στην οθόνη, η σημασία της χρηματοδότηση για το κάθε κράτος μέλος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ του, στον αριστερό άξονα, στον κατακόρυφο άξονα και κατά κεφαλή στην Ευρώπη, στον οριζόντιο, μας δείχνει μια σημαντική διακύμανση της οικονομικής σημασίας των πιστώσεων για την κάθε χώρα. Που δεν αντιστοιχεί σε επίπεδο εφημερίας οφειλόμενα στο μηχανισμό των ε, πιστώσεων. Και με τα σημεία αυτά, τα εισαγωγικά, θα ήθελα να περάσω στις, στους θεματικούς τομείς, στους οποίους κατευθύνονται οι πιστώσεις. Οι περισσότερες, όπως βλέπετε, είναι στο πράσινο, στις πράσινες γραμμές, δηλαδή υποδομές, σιδηροδρόμους, οδικά δίκτυα, ναι. λοιπές μεταφορές, ευρυζωνικές επικοινωνίες περιβάλλων ναι. και σε χαμηλότερο βαθμό στη γνώση και καινοτομία ή στην κατάρτιση και την εκπαίδευση. Τώρα ως προς την, ε, τις ε, επιδόσεις. Ενδιαφέρον να κοιτάξουμε αναδρομικά την περίοδο 2004-2006 παραδείγματι όπου έχει κλείσει ένας ολόκληρος κύκλος δαπανών και βλέπουμε ότι είχαν καλά αποτελέσματα οι ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τις επιδόσεις τους και συγκρινόμενες με το μέσο όρο των 25 της Ένωσης. Στην πρώτη περίοδο δηλαδή, με την ε, χρηματοδότηση των Ταμείων Συνοχής έχουμε μια μεγάλη πρόκληση για τις χώρες, θα διαχειριστούν τα κονδύλια, αλλά και στην απορρόφηση και στην ε, απελευθέρωση κονδυλίων και στις ε, διορθώσεις είναι τα ποσοστά σχετικά καλά για τις χώρες για τις 10 ε, πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, συγκρινόμενα ειδικά με τα 25 της συνολικής τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2007 με 2013 δείχνει διαφορετική εικόνα, πολύ πιο περιορισμένη χρηματοδότηση, πιο δύσκολες συνθήκες, η απορροφήση αναφέρθηκε διαρκετές φορές στη συζήτηση, δείχνει στοιχεία και είναι τα στοιχεία μας από τις αρχές του καλοκαιριού, δεν είναι τελείως επικαιροποιημένα, αλλά πάντως δείχνει τεράστιες διαφορές απορρόφησης μεταξύ κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αν δεν κοιτάξει κανείς τους ρυθμούς αλλαγής τα τελευταία χρόνια, θα διαπιστώσει σημαντικές αλλαγές στο ποσοστό στο ρυθμό αύξησης του ποσοστού απορρόφησης. Οι χώρες με τη χαμηλότερη απορρόφηση είναι και αυτές οι οποίες έχουν τους βραδύτερους ρυθμούς βελτίωσης της απορρόφησης. Το ζητούμενο βέβαια είναι τι γίνονται με αυτές τις επενδύσεις. Πολύ ενδιαφέρον σε αυτή εδώ η διαφάνεια που μας δείχνει τα στοιχεία από την μονάδα αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, από το δίκτυο αξιολόγησης, προσπαθεί να καταγράψει πιο συστηματικά τι αντίκτυπο έχουν τα διαφορετικά ταμεία και στο στην περιοχή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εκτιμήσεις ε, της δημιουργίας της συνεργασίας σε πλήρη απασχόληση για την περίοδο αυτή και εδώ, εάν δούμε τις 9.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην τσεχική δημοκρατία, σε σχέση με τα όσα είπε και ο αναπληρωτής υπουργό και τις 10.000 ε, θέσεις εργασίας, είναι πολύ διαφορετικά τα στοιχεία. Τα στοιχεία παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαφορές όταν τα δούμε ευθυγραμμισμένα στον τρόπο υπολογισμού για όλες τις χώρες με την ίδια μεθοδολογία. Και το πρόβλημα που βλέπουμε, το πρόβλημα που προκύπτει από τα τέτοια δεδομένα, είναι η μεγάλη διακύμανση στην ποιότητα των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν αυτά. Στην συνθετική παρουσίαση στρατηγικής έκθεσης που παρουσίασε φέτος η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής προσπάθησε να διατηρήσει μια διπλωματική παρουσίαση της κατάστασης στην ε, συνοπτική της επισκόπηση με τις συνέπειε βεβαίω προ την κινητικότητα και τη δυνατότητα να κάνει κανεί κρίσει για το τι έχει πει, κάθε ταμείο και η χρηματοδότηση. Πάντω έχουμε στοιχεία όχι μόνο για θέσεις εργασίας που είναι δύσκολο να προσμετρηθούν, αλλά και για, την, για το παραγόμενο προϊόν που ίσως είναι πιο απτό. Και εδώ έχω μια επιλογή περιλάβει σε αυτές τις δύο διαφάνειες των στοιχείων που μας, προσφέρουν, προσφέρει το δίκτυο αξιολόγηση για την περίοδο αυτή. Και εδώ σημαντικό είναι όχι να κοιτάξουμε μόνο τα στοιχεία προϊόντος αλλά και τις ε, συνέπειες για την οικοδόμηση θεσμών και ανάπτυξη διοικητικών δομών και δυναμικού ε, που μπορούν να προσφέρουν αυτές οι δαπάνες, αυτά τα κονδύλια. Η πολιτική της συνοχής λοιπόν έχει σε ορισμένες περιπτώσεις ε, παρουσιάσει σημαντική, σημαντικό έργο ως προς την ανάπτυξη και κυρίως να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση και την χρηματοδότηση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των προτινωμένων πολιτικών. Και εδώ περνώ στην ε, διαχείριση της χρηματοδότησης και προσπαθώ να δώσω κάποιες ιδέες γιατί παρουσιάζονται τις αποκλήσεις ως προς την εφαρμογή στα νέα κρατημέλη, όπως ονομάζονται, όπου πολλά έχουν να κάνουν με την ε, ποικίλη πρόοδο που σημειώνεται, ποικίλους ρυθμούς δηλαδή πρόοδου, ε, της εξόδου από τα λεγόμενα γραφειοκρατικά συστήματα σε συστήματα δημόσιας διαχείρισης όπως ονομάζονται τώρα και για να επανέλθω στα όσα είπε ο κ. Κούμπιακ η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με τις εδαφικές μεθόδους αλλά και οι ε, δομικές διαφορές που παραμένουν έχουν μεγάλη σημασία. από, τις, από την ομάδα των 15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουμε ήδη ότι χρειάζεται χρόνος για να φέρουν αποτελέσματα αυτές οι, αυτά τα προγράμματα, αυτή η χρηματοδότηση. Στα δεκρά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διαπιστώνουμε διαφορές ως προς τη στρατηγική, τη στόχευση των προγραμμάτων τους δικαιούχους. Πολλές φορές ε, θεωρούν ότι είναι δωρεές οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση στα προγράμματα αυτά και της επιλογής των σχεδίων που μερικές φορές γίνονται μόνο με όρους χρονικούς. Ποιος έκανε πρώτο συνέτηση. Έτσι ήταν μάλλον βραδία η ανάπτυξη μιας ε, αντίληψης ορθής διαχείρισης των κονδύλων αυτών στα κράτη από το 2004 και μετά. Ωστόσο σημειώνεται μια αλλαγή αντίληψης, ένα πιο εκλεπτισμένο ε, σχεδιασμό, συμμετοχή, επένδυση στην ε, παραγωγή έργου ή σχεδίων καλύτερα, δηλαδή εταιρικέ σχέσεις για την εξασφάλιση ενός καλού σχεδίου και καλύτερη επιλογή τελικά των πιο ποιοτικών προτάσεων και αντίστοιχα αξιολόγηση πιο αποτελεσματική. Ε, πάντως δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε μια ικανοποιητική κατάσταση. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι δεν είναι περιορισμένα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τα προγράμματα αυτά είναι, είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 28 κράτη-μέλη. αλλά για να αναφερθώ στην παρατήρηση του κυρίου Μποστινάρου και τη σταθερότητα. Τα προβλήματα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει συνδυασμό ή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων ε, και άρα γίνονται πολύ, αλλά πολλαπλασιάζονται οι έλεγχοι. Καθυστερήσει παρουσιάζονται μέχρι και πολιτικοποίηση των αποφάσεων για την ε, επιλογή των έργων. Καθίσατε δηλαδή πολιτική επιλογή πιο σημαντική από τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα έργα αυτά. Και για να συνοψίσω. διδάγματα σημαντικά για την ε, υλοποίηση στην προσεχή περίοδο είναι τα εξή. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούν τα προγράμματα να... Ε, πώς μπορούμε τα προγράμματα να διαχειριστούμε αποτελεσματικά για να εξυπηρετήσουμε τους στόχους. Πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε τον στόχο, το αποτέλεσμα και το πλαίσιο που θα είναι στραμμένο και αυτό στο αποτέλεσμα, με καλύτερη επίτευξη των στόχων της πολιτικής και άρα θα πρέπει να επενδύουμε περισσότερο στο διοικητικό δυναμικό, mm-hmm. να έχουμε επαρκείς και ποιοτικού πόρους ανθρώπινους και διαδικασίες απλουστευμένες και ευέλικτες. Και είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα της πολιτικής εξαρτάται από την ύπαρξη μιας ουσιαστικής ε, και καλής διοικητικής δομής. Και πρέπει να καταμετράται η, η διοίκηση έτσι ώστε να βλέπουμε ε, τα ουσιαστικά αποτελέσματα. Βέβαια, όταν η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης δεν είναι καλύτερη, όταν υπάρχουν ακόμη ελλείψεις προς το δυναμικό, μπορεί μια ποιοτική ηγετική στάση να αλλάξει αρκετά και να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Λαβέλτζου Γκαμπριέλ. Φρύπτου, που είναι Γενικός Διευθυντής ε, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη και συνοπτική παρουσίαση για μια εμπειρία από την Ρουμανία σε ό,τι αφορά την πολιτική για την ανάπτυξη και θα προσπαθήσω, όπως είπα, να το δυνατόν πιο σύντομο. Τρία βασικά θέματα μία μικρή παρουσίαση για τα καλά και κακά στοιχεία της πολιτικής, κάποια διδάγματα και κάποια συμπεράσματα. Βασικά η Ρουμανία αποτελείται από οκτώ αναπτυσσόμενες περιοχές χωρίς διοικητική ικανότητα στην παρούσα φάση, μάλλον στην φάση που ξεκίνησε η πολιτική. Και Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αστικών κέντρων, ε, κάποια, πόλη ανάπτυξη και 13 ε, κέντρα αστικής ανάπτυξης πέρα από το, πρωτεύουσα. Αυτά που είναι σημαντικά για τα κέντρα αυτά είναι τα προγράμματα που δίδουν πόρους και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη κέντρων ανάπτυξης, βελτίωση των υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και ανάπτυξης των κέντρων επιχειρηματικότητας. Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, 13,5% του συνολικού προγράμματος, τα αναπτυσσόμενα ε, κέντρα, λάβαν περίπου 6% συνολικά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποια θετικά χαρακτηριστικά για την πολιτική για τους πόλους ανάπτυξης. Καταρχάς, ε, μια σαφή, ένα σαφής εντοπισμός των ε, πόλων αυτών. Μιλάμε λοιπόν για κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη της, όλης της χώρας. Ύστερα, ένας πόλος ανάπτυξης αναπεριφέρεια για να ενθαρρυνθεί η ισόρροπη, βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Και σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των αστικών περιοχών στις ε, γειτονικές περιοχές. Και τρίτον, αυτό το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση τους έχει να κάνει με τις πόλεις που δημιουργούν μητροπολιτικές περιοχές και προετοιμάζουν ενωπημένα σχέδια ανάπτυξης. Τώρα, κάποια προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την πολιτική αυτή. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σαφής κατανόηση για το πόσο ο σχεδιασμός των πόλων αυτών μπορεί να συμβάλλει στη γενική ανάπτυξη της χώρας. Επίσης ε, βασίζεται σε περιφερειακά σύνορα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες συνέργειες. Επίσης, οι περιοχές ανάλυσης και παρέμβασης είναι περιορισμένες συνήθως. 30 χιλιόμετρα συνήθως γύρω από τις πόλεις. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, συμπερίληψη άλλων λειτουργικών οικονομικών περιοχών. Οι πιο μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές ε, δίνουν καλύτερες κίνητρα για επενδύσεις. Τέλος, η δημιουργία μητροπολιτικών περιοχών βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε συμφωνίες μεταξύ των τοπικών αρχών. Αυτό στην πράξη δημιουργεί σε δημιουργία ενώσεων και ενός, αν θέλετε, και περιοχών που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των λειτουργικών περιοχών. Κάποια διδάγματα από το παρελθόν τώρα. Οι οικονομικές αρχές διδάσκουν ότι σε κάποιες πόλεις είναι πιο μεγάλη, στις πόλεις είναι πιο μεγάλη ανάπτυξη και ότι χρειάζεται δημόσια επένδυση, αλλά και σε πιο χαμηλής ανάπτυξης περιοχές στην πράξη για το μέλλον της πολιτικής ανάπτυξης, θεωρούμε ότι έχουμε μάθει το εξής μάθημα. Ανάλυση του περιφερειακού ορίου μέχρι του οποίου υπάρχει σαφής αντίκτυπος. Καλύτερη και πιο στοχευμένη παρέμβαση βάσει το συγκεκριμένο σύνολο των ιδιαιτεροτήτων των πόλων αυτό το όριο των 30 χιλιόμετρων προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά. Χρειάζεται λοιπόν να προβλέψουμε μια ανάπτυξη των πόλων αυτών. Τώρα. Τα πραγματικά αναποιημένα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσεως με κατάλογο προγραμμάτων και τη χρηματοδότησή τους και από τον Εθνικό ενδεχομένω και Περιφερειακό Προπολογισμό. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να εξετάσει ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχουν οι Μητροπολιτικές Περιοχές και πώς μπορούν να, δημιουργηθούν, να συνέργειες. Και στο πλαίσιο αυτό, αυτή η επένδυση και σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να γίνει με τη σωστή χρηματοδότηση. Ένα άλλο πρόβλημα έχει να κάνει με το σχεδιασμό και το μηχανισμό υποπτίας και αξιολόγησης. Θα πρέπει να βρούμε τους σωστούς δείκτες. Είναι κρίσιμο αυτό για τον καλό σχεδιασμό της πολιτικής αυτής, αλλά και για την παρακολούθηση της απόδοσης της πολιτικής. Οι δείκτες αυτές θα πρέπει να είναι εύκολοι στην συλλογή και στην ερμηνεία. Άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Η δομή για τους πόλους ε, ανάπτυξης τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίε που διαχειρίζονται τους πόλους ανάπτυξης θα πρέπει να συμπεριλάβουν και τις δύο δομές που εκπροσωπούν τις κοινότητες αλλά κινητοποιώντας και τις τοπικές κοινωνίες. Με υποστηρίξη απόλυτα επίπεδα και θα πρέπει να δοθεί πιο πολύ σημασία στην ανάπτυξη δυναμικού, στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί τέτοιου είδους θεσμούς. Και τέλος, να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη, καλύτερη ε, σχέση μεταξύ των πολιτικών, γιατί α, οι πόλοι ουσιαστικά αποτελούν κινητήριο δύναμη για την χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πολιτική οικονομικής ανάπτυξης, η οποία θα συμβαδίζει και στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορεί να συμπληρώσει τις πολιτικές αυτές, δίδοντας τους μηχανισμούς και βελτιώνοντα το επιχειρησιακό περιβάλλον σε ό,τι αφορά τους πόλους αυτούς και κάποια συμπεράσματα. Η πολιτική για την ε, ανάπτυξη των πόλων και πώς θα συνεχιστεί. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την στρατηγική το 2020, μια δέσμευση για μια σωστή ανάπτυξη. Χρειάζονται κάποιες εμβληματικές πρωτοβουλίες και κάναμε κάποια σχόλια για το πώς οι ε, πόλοι ανάπτυξης μπορούν να συμβάλλουν στην επιτεύξη των στόχων αυτών. Δεν τονίζεται φυσικά στις πρωτοβουλίες αυτά σε ιδιαίτερο σε περιφερειακή διάσταση. Θεωρούμε ότι οι προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε για τους πόλους ανάπτυξης υποστηρίζουν τις πολιτικές αυτές. Για παράδειγμα, η Ρουμανία έχει Ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλλά αυτά βρίσκονται κυρίως στις μεγάλες πόλεις και μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα. Αυτό καταδεικνύει ότι σε ό,τι αφορά το Youth on the Move, σε ό,τι αφορά άλλες ε, πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης και αυτοί σχετίζονται με την πολιτική ανάπτυξη των πόλων και σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας Και η πρωτοβουλία για την αποδοτικότητα της ενέργειας τονίζει και τη διάσταση των μεταφορών, δίδοντας ειδικότερη έμφαση στην ε, διαφορετική χρήση και συνδυασμό τρόπων μεταφοράς. Μιλάμε για μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται. Και θεωρούμε λοιπόν ότι οι πολιτικές για την ανάπτυξη ε, των πόλων θα συνάδουν και θα συμβαδίζουν με την πολιτική το 2020. Τέλος, ε, οι πόλοι ανάπτυξης ε, μπορούν να υποδεχτούν τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, γιατί μιλάμε για μεγάλη οικονομική μάζα, όπου μπορούν να υποφεληθούν και οι ιδιωτικές εταιρείες και οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο και να δώσουν όθηση και στην ανάπτυξη αλλά και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της πολιτικής αυτής και την έχει συμπεριλάβει και στα νέα πακέτα. Για την περίοδο 2014-2020 και σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάπτυξη των αστικών κέντρων και καλεί τις χώρες να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή ιδανικά μια ενοποιημένη προσέγγιση δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο για να προσελκύει τους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά ως ένα εργαλείο για να υποστηρίξει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, που δεν θα πρέπει να υπονομεύεται, για παράδειγμα, ένα σύστημα μεταφορών σε μια μεγάλη πόλη μπορεί να προσελκύσει πόρους και μετά να καταληφθεί εφόσον τελειώσει αυτή η χρηματοδότηση. Άρα θα πρέπει οι πόροι αυτοί να εξυπηρετούν πιο γενικούς σκοπούς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Thank uh, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία όλα τώρα να μας κάνει τη δική της παρουσίαση. Άλντα Οζόλα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Άλντα και Οζόλα. Είμαι από τη Λετωνία και εκπροσωπώ εδώ μία μη κυβερνητική οργάνωση για όλες τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες που λέγεται CEE Bankwatch Network. Η παρουσίασή μου βασίζεται και στη δική μου εμπειρία στη χώρα μου αλλά και στην εμπειρία άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης. Βεβαίως αυτά που θα σας πω είναι από την άποψη της κοινωνίας των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι έχουμε αρκετή εμπειρία και εγώ προσωπικά παρακολουθώ την χρήση και απορρόφηση των ενωσιακών κονδυλίων εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε να κάνουμε μερικά σχόλια λοιπόν και για τα μαθήματα που μπορούν να δοθούν ή τις συμβουλές για την χρηματοδότηση από την Ένωση. Να σας δείξω μία γραφική παράσταση της Κομισιόν για να δείξουμε τη σημασία που έχει η ενωσιακή χρηματοδότηση στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Οι χώρες αριστερά αντιπροσωπεύουν το μερίδιο των ενωσιακών κονδυλίων στις συνολικές δημόσιες επενδύσεις. Βλέπουμε ότι στην κεντροανατολική Ευρώπη το μερίδιο αυτό είναι περίπου 50% και σε ορισμένες ακόμα ψηλότερο όπως στην Ουγγαρία και άλλες. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συγχρηματοδότηση αλλά μας ενδιαφέρει επίσης και η σωστή και αποτελεσματική χρήση των χρημάτων αυτών. Τώρα, μαθήματα από λάθη του παρελθόντος, για οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις τουλάχιστον, θεωρούν ότι, για να μην επαναλάβω θέματα που έχουν αναφερθεί από προηγούμενους, ότι οι χώρες μαθαίνουν από τα λάθη τους γιατί έγιναν πολλά λάθη, όχι επίτηδες βέβαια. Δήμοι και κοινότητες θέλησαν να επιδείξουν μεγαλύτερη ευελιξία για να προσαρμοστούν στις πραγματικές συνθήκες και καμιά φορά δήλωσαν δαπάνες ότι είναι ως απαράδεκτες. Και επίσης υπήρξε, σημειώθηκε και κάποια διαφθορά. Όλα αυτά βέβαια κόστησαν στο φορολογούμενο. Γιατί όταν κάνει λάθη ένας Δήμος ή μια κοινότητα, τα πληρώνει ο φορολογούμενος τα λάθη. Επίσης υπήρξαν, σημειώθηκαν γελία σχέδια και προγράμματα, όπως τεράστια στάδια που χτίστηκαν σε απομακρυσμένες περιφέρειες. Είναι μη ρεαλιστικά σχέδια αυτά και οι Δήμοι τα ζήτησαν απλώς και μόνο γιατί είχαν τα χρήματα. Υπάρχει λοιπόν μια έλλειψη στρατηγικής προσέγγισης εδώ και ελπίζω να μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα λάθη. Επίσης πιστεύουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις η σημασία της πολιτικής συνοχής πρέπει να εξηγείται καλύτερα στους πολίτες. Παραδείγματο χάρη συχνά σε επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, η συσχέτιση μεταξύ βελτίωσης της ποιότητας της ζωής δεν εξηγείται άμεσα από την πολιτική συνοχής, ενώ θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει ότι και αυτή συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, μερικές φορές δεν υπάρχει αρκετή συνέργεια ή συνεργασία. Θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων και από αυτό υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ας πούμε κάποιος δήμος ασφαλτώνει έναν δρόμο και μερικούς μήνες αργότερα από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα βάζουν σωλήνες νερού στον ίδιο δρόμο καταστρέφοντάς τον ταυτόχρονα και τέτοια πράγματα πρέπει να αποφεύγονται γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικά ή ωφέλιμα. Υπάρχουν όμως και θετικά σημεία. Να σας εξηγήσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, πολύ θετικό για την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας σε μια πολυκατοικία. Όταν άρχισε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν πολύ δημοφιλές, αλλά μετά, επειδή το πήραν πολύ σοβαρά η κυβέρνηση και το Υπουργείο, έγινε μια μεγάλη καμπάνια πληροφόρησης και χαλαρώθηκαν πολλοί γραφειοκρατικοί κανόνες και τελικά έγινε πολύ δημοφιλές το πρόγραμμα και μείωσε κάπως τον αντίκτυπο της σκληρής οικονομικής κρίσης και δημιούργησε και θέσεις εργασίας και το περιβάλλον. Σε άλλες χώρες επίσης έχουν σημειωθεί τέτοιες θετικές εμπειρίες. Αυτή όμως η δικιά μας ήταν πολύ θετική. Και αυτό σημαίνει ότι αν ένα πρόγραμμα δεν είναι δημοφιλές από την αρχή πρέπει να γίνουν προσπάθειες να εξηγηθεί Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω μερικά μικρά προγράμματα για τους πολιτικούς βέβαια η προώθηση των μεγάλων σχεδίων είναι αυτό που τους ενδιαφέρει γιατί αυτά είναι πιο ορατά και είναι πιο εύκολο να επιδειχθούν στους εκλογίστους ως επιτεύγματα, αλλά και τα μικρά προγράμματα μπορεί να είναι ωφέλιμα και να συνεισφέρουν και αυτά στην κοινωνική συνοχή. Ας πούμε τα προγράμματα τύπου Leader, όπου διάφοροι ενδιαφερόμενοι συνεργάζονται και σχεδιάζουν στρατηγικά την τοπική οικονομική τους ανάπτυξη. δεν θα σας επαναλάβω ποια είναι η κίνδυνη των μεγάλων προγραμμάτων γιατί ακούσαμε προηγουμένως ότι τα μεγάλα προγράμματα έχουν περισσότερους κινδύνους διαφουθοράς και καθυστερήσεων. Ποιες είναι οι προοπτικές λοιπόν και οι προτεραιότητες μας για την περίοδο 14 με 20. Τρεις. Πρώτον οι εταιρικέ σχέσεις. Το είπαν και άλλοι αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, έχει βελτιωθεί σε μερικές χώρες περισσότερο από τις άλλες, αλλά πιστεύουμε, εννοούμε όταν λέμε εταιρική σχέση, εννοούμε τις τοπικές αρχές, κοινωνικούς εταίρους και μη κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορούσαν αυτά όλα η τέτοια συνέργεια να βελτιώσει τα προγράμματα και να αποφευχθούν διάφοροι κίνδυνοι, ιδίω ήδη από την φάση του σχεδιασμού και με προσέγγιση περισσότερο στοχευμένη στα αποτελέσματα. Όχι μόνο όμως στο σχεδιασμό αλλά και στην εφαρμογή. Εδώ οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι τοπικές αρχές καθώς και άλλοι παράγοντες θα έπρεπε να αντιπροσωπεύονται περισσότερο και καλύτερα για την εποπτεία της χρήσης των ενωσιακών κονδυλίων. Γιατί η παρουσία τους συμβάλλει περισσότερο στην ε, αίσθηση της κοινωνίας ότι το πρόγραμμα τους ανήκει. Επίσης θα θέλαμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σας είπα ήδη για τα προγράμματα τύπου Leader. καθώς και την τοπική ανάπτυξη με βάση τις κοινότητες. Δυστυχώς πολύ λίγες χώρες το χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο προγράμματος με τα αρχικά CLDD. Η Σλοβακία είναι καλό παράδειγμα. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης των τοπικών αναγκών, να δοθεί περισσότερο, να δοθούν περισσότερες δικαιοδοσίες στις τοπικές αρχές. Για γιατί αυτές είναι εκείνες που ξέρουν καλύτερα ποιες είναι οι, ανα, τοπικές ανάγκες και είναι και σε θέση να εφαρμόσουν σε καλύτερο χρονοδιάγραμμα τα πράγματα είπα πριν ο ένας να ασφαλτώνει το δρόμο και ο άλλος να τον ξανασκάβει για να βάλει σωλήνε. Τονίσανε και άλλοι ότι στη νέα προγραμματική περίοδο η προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα είναι η καινούργια βάση. Ακόμα δεν το έχουμε δει βέβαια. Ίσως να εφαρμοστεί στις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει. Η ενδυνάμωση των οριζοντίων αρχών, μεταξύ των οποίων το περιβάλλον, η βιωσιμότητά του δηλαδή, πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα. Και τέλος, θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να είναι συνεπής και όχι αντίθετη με άλλα ενωσιακά προγράμματα όπως τα κλιματολογικά και τα περιβαλλοντολογικά. Επίσης το Ένωση 2020 δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τα προγράμματα της συνοχής. Μερικές φορές δεν υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλίδες. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις το παρακολουθούν αυτό στενά. Και ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Μερικές φορές επίσης είδαμε ότι υπάρχουν οι σωστές εκφράσεις και διατύπωση και ορολογία Δυστυχώς όμως μερικές άλλες φορές η ορολογία αυτή είναι απλώς μια κάλυψη γιατί ας πούμε όλα δεν είναι χρήσιμες όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το περιβάλλον καθώς και η προσαρμογή στην αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών δεν γίνεται πάντοτε με τον τρόπο που πρέπει, γίνεται διακοσμητικά ή σαν διασκέδαση. Αυτά τα παρακολουθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Βαλεντόφσκι τώρα. Από το Τεκνόπολης Group Belgium. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Κυρίε και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το μικρόφωνο του ομιλητή δεν είναι αναμένο. Δεν είναι αναμένο. Το μικρόφωνο του ομιλητή δεν ακούγεται. Ο μιλητής δεν ακούγεται. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα λοιπόν να φερθώ στα διευθυντικά ταμεία και την εμπειρία μας από τις παρεμβάσεις και την έρευνα που έχουμε κάνει. Θα ήθελα να δώσω κάποιες βασικές παρατηρήσεις καταρχάς, ίσως για να δώσω όθηση, βάση για συζήτηση και ίσως να απαντήσω σε κάποια ζητήματα τα οποία ίσως δεν μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε πλήρως, δηλαδή τι είδους αντίκτυπο έχει η πολιτική αυτή της καινοτομίας ερωτικά ταμεία. Δεν μιλούμε λοιπόν μόνο για ένα είδους έρευνας, είμαστε συντονιστές από τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακής Πολιτικής και παρακολουθούμε σε 200 περιφέρειες την ε, καινοτομία. Εδώ και 13 χρόνια μάλιστα κάνω αυτή τη δουλειά εγώ. και παρακολουθώ την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η έρευνα, τα, προγράμματα που απευθύνονται σε υποδομές έρευνας, εργαστήρια, κτίρια ή την ίδια την έρευνα αυτή καθεαυτή είναι τα κύρια έργα που υποστηρίζονται, υποστήριξη προς τις εταιρείες συνήθως στοχεύει σε μεμονωμένους δικαιούχους, μεμονωμένες εταιρείε δηλαδή, σε σχέση με πιο προηγμένες οικονομίες που χρειάζονται πιο περίπλοκα μέτρα και ενσωμάτωση και σύμπραξη διαφορών εταιρείων. Βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα εδώ, δηλαδή με μονομένους δικαιούχους. Επίσης, βλέπουμε μια τάση μίμησης πολιτικών σε διάφορες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες του, των τύπων ε, των μέσων. Αυτά στόχο έχουν όχι μόνο να βελτιώσουν ε, τη διακυβέρνηση αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για την καινοτομία και την εισαγωγή πολιτικών ε, στόχευμένων στην καινοτομία. πέραν της ανταπόκρισης στις πολιτικές, αν περάσουμε στη διαχείριση, στην διοίκηση, πολλά ακόμα μένουν να γίνουν. Τα σχετικά συμβούλια δεν φαίνεται να παίζουν το ρόλο που θα όφυλαν. Υπάρχουν εμπόδια στην ε, υλοποίηση και διαφορετικές ερμηνείες ακόμη σε εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας, δηλαδή το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε βέβαια και ένα πλέγμα μέτρων πολιτικής δάνεια ή τύποι εγγυήσεων που προβλέπονται, που μπορεί να περιπλέκουν και να δυσκολεύουν ε, την ε, ροή των προγραμμάτων. Και θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω εδώ ότι στην αναζήτηση μιας ενός κατακόρυφου συντονισμού με ένα κεντρικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καλύτερος τρόπος για την κατανομή των ε, ευθυνών και της χρηματοδότησης είναι ο στόχος στον οποίο ε, αποδίονται τώρα οι διαπραγματεύσεις ορισμένες τουλάχιστον χώρες. Και όταν μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για θεματική συγκέντρωση, εξειδίκευση, και ούτω καθεξής. Από τις χώρες και Ανατολικής Ευρώπης βλέπουμε ότι ξεκίνησε με αυτή η προσπάθεια, αλλά οι μεθοδολογίες ήταν μάλλον παραδοσιακού τύπου. Και άρα χρειάζεται βελτίωση στην εξειδίκευση και τον εξεχρονισμό. Το να δούμε τώρα πώς αλλάζουν αυτές οι πολιτικές καινοτομίες, την περιφερειακή καινοτομία και τα συστήματα περιφερειακής καινοτομίας στην Ευρώπη. Εδώ βλέπετε τον πίνακα βαθμολογίας της περιφερειακής καινοτομίας, μια στατιστική ανάλυση των στοιχείων που έχουμε στη θέσή μας και δεξιά το monitor, την ε, παρακολούθηση της περιφερειακής καινοτομίας που έχει αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση αναπτύξει. Και εδώ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε και να αναλύσουμε την ε, κίνηση και τις συνέπειες των πολιτικών που καταγράφει το δίκτυο των περίπου 100 ανταποκριτών που έχουμε στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Δίνω λοιπόν κάποιες εικόνες εδώ δαπανών από την έρευνα και ανάπτυξη με τα 15 πρώτα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρχάς. που δείχνουν 160 δις ευρώ, Φερρυπίν, για ορισμένα κράτη-μέλη με χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη των 12. Οι τάσεις μπορεί να φαίνονται αυξητικές, βλέπουμε όμως σε σχέση με τις δαπάνε αν επιχείρηση για έρευνα και ανάπτυξη από το 95 και στα δεξιά βλέπετε τους 12, Ευρώπη των 12, με 45 έως και 50% των επιχειρήσεων στην έρευνα και ανάπτυξη. Μια εικόνα όμως που παραμένει χωρίς σημαντικές αλλαγές. Και αν κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες, που δεν έχω αυτή τη στιγμή το χρόνο να σας εξηγήσω, αν κοιτάξουμε πιο διαρθρωτικούς μακροπρόθεσμους δείκτες, δεν παρουσιάζονται σημαντικές αλλαγές για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αν δείτε δηλαδή τα μεγέθη των επιχειρήσεων που επενδύουν στην κοινοτομία στην πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι αυτό. Τώρα τι ξέρουμε για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής, των επιλεγόμενων πολιτικών. Οι τελευταίες δύο προτεραιότητες που υπογραμμίζονται εδώ, αναφέρουμε και εξηγούμε ότι έχουν θετικό αντίκτυπο και αποτέλεσμα και έχουμε τις δύο πρώτες κατηγορίες εδώ με επίκριση ότι είναι πολύ νωρίς ε, για να δώσουν μια αξιολόγηση για το μέτρο ή ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση αλλά χωρίς πιο συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την επίτευξη του στόχου. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι η αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής ακόμη δεν είναι γνωστό εάν έχει φέρει αποτελέσματα, δεν υπάρχει η θετική αξιολόγηση ακόμη στο βαθμό που θα θέλαμε. Και εδώ με αυτή τη διαφάνεια θέλω να συγκρίνω με τα στατιστικά δεδομένα αναπεριφέρεια τις πολιτικές και την αποτελεσματικότητά τους και εδώ προσπαθώ να δείξω πιο θετικές αξιολογήσεις της θεματολογίας και των πολιτικών περιφερειακής καινοτομίας που είναι πιο θετικές πάντα στις ε, περιοχές εκείνες που έχουν γενικά καλύτερη κατάσταση, που έχουν ηγετική θέση. Και μετά, όπως βλέπετε, ευθύνουν τα ποσοστά, ανάλογα με την περιοχή και, τη, και η θετική ανταπόκριση. Κύρια μηνύματα λοιπόν, ότι παραμένει μια σημαντική πρόκληση το να κλείσει το χάσμα καινοτομία μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Δεύτερον, ότι μπορούν οι αποτελεσματικές πολιτικές να φέρουν μια σημαντική διαφορά και ότι είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, την πορεία μιας περιφέρειας. Εδώ λοιπόν αναφερόμαστε σε μέτρα για τις 200 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτουμε και τα οποία έχουμε καταμετρήσει, αλλά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει γραμμική σχέση αιτιότητας, αλλά ότι μπορούμε κάποιες επιδόσεις προς την καινοτομία να τις εξηγήσουμε χάρη σε αυτές τα μέτρα. Δηλαδή για κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα οι πιο καινοτόμες περιφέρειες έχουν εισαγάγει τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο τέτοιου είδους μέτρα. Καινοτομία λοιπόν και το πιο σημαντικό είναι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση στη διακυβέρνηση, περισσότερη ευελιξία, διάθεση για ανάληψη κινδύνου, αλλά και πιο ευέλικτη προσέγγιση διαχείριση στη διακυβέρνηση και βέβαια προσεκτική επιλογή των κριτηρίων διαλογής από τις υπηρεσίες αξιολόγησης καθώς και ενδεχομένως ένας φορέας ο οποίος θα ασχολείται με την αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων αυτών, ώστε να κατευθύνονται αυτά προς την καλύτερη δυνατή κατεύθυνση και βέβαια τελευταία παρατήρηση, υπάρχει περιθώριο για βελτίωση της αξιολόγησης και του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα εντάσσονται μέσα στις δικασίες εκμάθησης. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε στοιχεία βεβαίω εδώ για το Τεχνόπολη όποτε θέλετε και αν είστε σε ένα προσεχέ εργαστήριο. Σα ευχαριστώ κύριε Κυρίλοφ, είναι ο πρώτο ομιλητή. Ε, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Μία ερώτηση έχω να κάνω που δεν είναι απλή ασφαλώ, δεν είναι απλή στην απάντησή τη. Είναι ένα θέμα για συζήτηση μάλλον προς την κυρία Οζόλα και στον καθηγητή Μπάχτλερ. Ασφαλώς υπάρχουν ε, διαφόρων ειδών διοικητικές δομές στις χώρες μας. Και φυσικά υπάρχει διαφορετική προσέγγιση κεντρική, κεντρική διαχείριση ως μέθοδος εργασίας, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε προβλήματα συντονισμού. Αυτό έχει ήδη αναφερθεί. Ίσως με τις, λιγότερο, με τις πιο μικρές χώρες, μία ενιαία υπηρεσία, μία προσέγγιση μπορεί να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ το έχω δει προσωπικά αυτό στην Εστονία, όπου μία υπηρεσία μπορεί να λάβει τέτοιες εργασίες. Ασφαλώς αυτό είναι πιο δύσκολο για μεγάλες χώρες. Να σας ρωτήσω όμως, Υπάρχουν άλλα παραδείγματα από τις χώρες σας, από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, από τις νέες χώρες μέλη, που καταδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο αυτών μοντέλων. Ευχαριστώ, Ευγένη. Να πω, λέει η Πρόεδρος, ότι έχουμε 5-6 ομιλητές ακόμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για τον καθένα σας, για εκτενέστερα σχόλια σας. Παρακαλώ, σύντομα σχόλια και ερωτήσεις να κάνετε. Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να απευθυνθώ στον καθηγητή Μπάχτλερ να τον ευχαριστήσω γιατί προσυπογράφεται και επιβεβαιώνεται αυτά που είπα για τη Ρουμανία, δυστυχώς. Δύο στοιχεία προς τον Ρουμάνο ομιλητή, τον κύριο Φρύπτου. Καταρχάς, είναι σαφές μετά το θέμα που παρουσιάσατε ότι η πόλη είναι το καλύτερο επίπεδο να ε, εφαρμοστεί αυτή η πολυταμιακή και πολυεπιπεδή προσέγγιση. Πώς προετοιμάζει η Ρουμανία το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής και την σχετική εφαρμογή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι από τα διάφορα ταμεία αλλά και αυτή η συνολική προσέγγιση. Κατά δεύτερον, πώς θα διαχειριστούμε τα project πολλαπλών ταμείων, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την εφιστάμενη υποδομή η Ρουμανία θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Τι θα κάνουμε και πότε. Αν δεν ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο του 2014, κάποια άλλη μετέπειτα χρονική στιγμή, προκειμένου να αγγίθουμε μια επιτυχή εφαρμογή. Και ένα τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά τους πόλους ανάπτυξης. Το ξέρω καλά, την ξέρω καλά αυτή την ιστορία, αλλά αυτό που κρύβεται από πίσω δεν είναι τόσο ευτυχές. Καταρχάς, η διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν ήταν τόσο δημοκρατική. Λίγο λόγο είχαν άλλοι φορείς πέρα από τις μεγάλες πόλεις. Και κατά δεύτερον, ακόμα απουσιάζει μία στρατηγική αστικής ανάπτυξης και μία στρατηγική ενέργειας στη χώρα μου, γιατί οποιαδήποτε αστική ανάπτυξη σχετίζεται τουλάχιστον με μία στρατηγική αστικής ανάπτυξης και μία στρατηγική ενέργειας. Αυτά συμβαδίζουν το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ, κύριος Γκουτμάνης. Εγώ μία μικρή ερώτηση έχω να κάνω προς τον ε, από ε, της Ρουμανίας. Ακούσαμε τις φήμες που λένε ότι άλλαξαν τα συστήματα ελέγχου ανεξάρτητα. Τα αλλάξατε χωρίς να γίνουν αυτά αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως αυτό είναι ο λόγος που υστερείται τόσο πολύ σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που έχει να κάνει με την απορρόφηση σε ό,τι αφορά και την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σόλμπριχτ. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση να κάνω. Μία τεχνική φύσεως παρατήρηση να ζητήσω από τη γραμματεία να ενημερώσω στο μέλλον του ομιλητέ ότι έχουμε μικρέ ε, οθόνες και ε. δεν μπορούμε να διαβάσουμε τι εμφάνισε αυτέ που προορίζονται για μεγάλε ε, οθόνες. Δεν ξέρω τι είναι και θέμα ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό δεν έχουμε πάντα μεγάλες οθόνες. Κάποιες φορές έχουμε μικρές οθόνες. Άρα σας παρακαλώ στείλτε μας και τις παρουσιάσεις μετά την ε, συνάντηση. Θα μας βοηθούσε ιδιαίτερος. Μία ερώτηση να κάνω και όποιος θέλει να απαντήσει. Ίσως να τη θέσω πρώτα στον Τζον. Όντως, οι κατηγορίες που έχουν οριστεί ακόμα στην Ευρώπη ισχύουν. Η αναλυτική κατηγορία είναι αυτή που μετράει. Η πολιτική κατηγορία είναι χρήσιμα σε αυτά. Σήμερα έχουμε την κεντροανατολική Ευρώπη, τι νέε χώρε. Αυτό είναι πολιτική κατηγορία. Εμεί πίσω από το τέχος του Μερολίνου είμαστε καινούργιε. Δεν έχουμε πει ποτέ ότι η Μάλτα ή η Κύπρος είναι καινούργιε χώρε, μέλη. Έχουμε την κεντροανατολική Ευρώπη, τα νέα κράτη-μέλη, του στην Ευρώπη των 15. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσον υπάρχουν ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένα για τις ε, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης από την έρευνα. Οι διαφορές, για παράδειγμα, μεταξύ της χύψη χώρας και της Ελλάδας, της Πορτογαλίας. Είναι ένα θέμα αυτό που έχει τεθεί, δεν έχει τεθεί από την Επιτροπή, αλλά υπάρχει πραγματικά τέτοιος λόγος ανάλυσης κατηγοροποίησης Ευχαριστώ. Να πω στο Γιάννη λέει πρόεδρο ότι εγώ ακούω κάποια πράγματα που δεν τα ακούτε απαραίτητα εσείς. Αν μιλάει κάποιος ε, από την Ευρώπη των 15, κανείς δεν μιλάει για τις χώρες μας, αλλά σήμερα όλοι μιλούν για τις χώρες μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ταυτότητα που τη δημιουργούμε εμείς και την επιβάλλουμε στους υπόλοιπους. Εμείς αισθανόμαστε σαν ένα σύνολο εμείς μιλάμε για το σύνολο των χωρών μας. Ο κύριος Νίλσεν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ειδικά. Θα μιλήσω λοιπόν σου ειδικά. για να είναι βέβαιο ότι αυτά που λέω μεταφράζονται και γίνονται κατανοητά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω τις εμπειρίες άλλων και υποφελούμε από αυτές ως προς τις ανάγκες που θα έχουμε στο μέλλον. Αυτό που χρειάζομαστε είναι η ειλικρίνεια και τιμιότητα. Δεν αρκεί να συναντιόμαστε με ένα μικρό με αριθμό ανθρώπων. Χρειαζόμαστε ευρύτερο κυκλοφωνών που ακούμε. Με μεγάλη χαρά άκουσα για την εμπειρία της Λετωνίας γιατί εδώ βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι οι εταιρικές σχέσεις. Έτσι μας είπε η εκπρόσωπος της και το βρίσκω πολύ σωστό. Στην Επιτροπή μας έχουμε διαπιστώσει ότι η εταιρική αρχή είναι η βάση του μέλλοντος. Πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι παράγοντες να συνεργάζονται σε ένα πρόγραμμα και στο σχεδιασμό του ήδη γιατί μόνο έτσι γνωρίζει κανείς όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται τοπικά με το πρόγραμμα και αν χρειάζεται μπορεί και να τους διδάξει πώς να το κάνουν καλύτερα. Εγώ το έχω ζήσει αυτό, ήμουν δήμαρχος μιας κοινότητας στη Σουηδία την στιγμή μέχρι να μπούμε στην Ένωση και δεν πρέπει να περιμένει κανείς να προσκληθεί σε διάφορες εκδηλώσεις. Πρέπει να κάνει αγώνα για να συμμετάσχει. Γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι στα κράτη-μέλη υπεύθυνοι και εκπρόσωποι της κυβέρνησης που θεωρούν ότι τα ξέρουν καλύτερα από σένα. Ο Ιωακίμ Τσέλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους σα ομιλητές για τις, απόψεις και τις αναλύσεις τους. Η διευθυντική πολιτική για τη συνοχή θα πρέπει να χρησιμεύει στην υποστήριξη των ε, πιο αδύναμων περιοχών στην Ευρώπη και τη δυνατότητα να καλύπτουν την υποχώρηση του, το, κενό που τις χωρίζει από τις προηγούμενες περιοχές. Αυτό είναι και το νόημα της τελευταία Πολιτικής Συνοχής. Και βλέπουμε ότι σε αρκετές περιοχές, παρότι έχουν διατεθεί πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, δεν έχει καλυφθεί το σχετικό κενό. Και μάλιστα μερικές φορές τελευταία ερχονται τα ταμεία αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση στοχεύσεων κυβερνητικών και μάλιστα με πολύ, κεντρική, με πολύ κεντρικό σχεδιασμό. Κυρίως υποδομές, οδικούς κόμβους κτλ. Για λόγους και με βιωσιμότητα που δεν αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον εγώ. Τα κράτη λοιπόν της Κεντρικής Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης διερωτώ με έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους μήπως ε, δεν έχουν δει ξεκάθαρα την κατάσταση και θα ήθελα έστω για το επιχείρημα, για να δεχθώ το επιχείρημα, να, να παραδεχθώ ότι έχουν ε, κατασκευαστεί έργα σημαντικά, καθαρισμού λιμάτων και το καθεξής χρήσιμα έργα. Αλλά εάν πια έχουν όλες οι πόλεις κέντρα καθαρισμού λιμάτων, τι άλλο μπορεί να χρειάζονται. Γιατί βέβαια η γερμανική επιχείρηση θα είναι αυτή η οποία θα κάνει τη σχετική, ε, τη σχετική κατασκευή, αλλά ε, πέραν το ότι βέβαια θα χαρεί πολύ να εισπράξει άλλα 70 δισεκατομμύρια, ε, δεν καταλαβαίνω σε τι μπορεί να εξυπηρετήσει να φτιάχνουμε και άλλες υποδομές στο ίδιο, στον ίδιο τομέα. Τα προβλήματα λοιπόν, τα οποία περιγράψατε σε ένα βαθμό κομψά, ε, φοβούμαι ότι δεν θα έχουν λυθεί και στην επόμενη περίοδο και προς το τέλος θα ξανασυστούμε γιατί θα είναι ακόμα πιο έντονα. Και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και για υποστήριξη της ευρωπαϊκής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και της παρουσίας της διεθνής αγορές. Ερωτώ λοιπόν, ποια είναι η δική σας προσωπική ανάλυση, που νομίζετε ότι μπορούμε να δώσουμε ε, έμφαση σε τι μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό. Το να πηγαίνουν τα κονδύλια μεταξύ άλλων σε ένα, σε ένα καλύτερο συντονισμό ουσιαστικά, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, και να μην χτίζονται μονοδρόμοι. Και τουλάχιστον αν χτίζονται να ξέρουμε ότι τους χρειάζονται και όλα κάτι και τις περιοχές. Πράγμα το οποίο σημαίνει και αηφορία και διασύνδεση με την αντίστοιχη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, τη σημασία για την περιοχή και το καθεξής. Για την επιστημονική έρευνα και καινοτομία με παραγωγή θα ήταν καλό πιστεύω να υπάρχει. Δυστυχώς όμως και στα κράτη κεντρική και ανατολική Ευρώπης η κατάσταση είναι μάλλον αργή, η εξέλιξη είναι μάλλον αργή και δεν ε, βλέπουμε αρκετή πρόοδο. Να μιλήσω κι εγώ και να ζητήσω από τον κύριο Λεβαντόσκι να πάρει το λόγο. Μάλλον αυτό που είπε ο κύριος Λεβαντόσκι σε ό,τι αφορά ε, την κοινοτομία που αποτελεί απόρρια των μεμονωμένων επιχειρήσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση με την έλλειψη μη κοινωνικού κεφαλαίου ή επίσης με την ε, παράδοση ιεραρχίας στην κοινωνία και στην οικονομία. Κινούμαστε προς μια διαφορετική κατάθεση. Θα ήθελα να σας δώσω λοιπόν το λόγο. Ποιος θα θέλει να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Τζον, θα θέλετε να ξεκινήσετε. Και στη συνέχεια, αν θέλει να πάρει το λόγο και η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Να επιλέξω αυτές, όχι τις εύκολες, αλλά επαστρεπτώσει αυτές που μου απευθύνθηκαν σε μένα. Ο κύριος Κυρίλοφ. Για το πώς προσμετρούνται οι διοικητικές ικανότητες. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα αυτό. Πολλά γίνονται από την Γενική Διεύθυνση Ρέτσι και Employment. Αυτό μας βοηθάει. Ωστόσο, εξετάσαμε κάποια στοιχεία. Καταρχάς η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και πώς ε, διαχειριζόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό, τις ε, ικανότητες, τις δομές, τη σταθερότητα, αλλά το επίπεδο διαδικασίας εκμάθησης, δηλαδή μια προσαρμογή μετά από τις εμπειρίες που συλλέγονται. Η αστάθεια ασφαλώς τα, τα διακόπτει αυτά και υπάρχει και το θέμα φυσικά της γενικότερης ε, κουλτούρας. Υπάρχουν ωστόσο κάποια στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι μικρότερες χώρες τα πηγαίνουν καλύτερα. σε ό,τι αφορά την απόδοσή τους και τις δυνατότητές τους. Στο Ίδρυμά μας κοιτάξαμε την περίοδο 2004 μέχρι 2008 και είδαμε ότι η διοικητική ικανότητα Εστονία, Λετωνία και Πολωνία ήταν οι καλύτερες χώρες σε ό,τι αφορά την ε, απόδοση αυτή. Αυτό δεν συνάδει με τη θεωρία μικρών και μεγάλων χωρών, αλλά και τότε ακόμα υπήρχε αποκέντρωση μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών. Σημαντική. Και η Ιστονία και η Λιθουανία σε ό,τι αφορά τα θέματα ικανοτήτων ήταν οι καλύτερε. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία που υποδεικνύουν αυτό που λέτε, αν και όχι ακόμα τεκμηριωμένα. Τώρα, αυτό που είπε ο Γιάννα Όλμπριχτ για την ε, κατηγοριοποίηση και κατά πόσο ισχύει αυτή η κατηγοριοποίηση. Κοιτάξτε, υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτή την κατηγοριοποίηση, ιδιαίτερα επειδή η ανάπτυξη προέρχεται και από την ε, πολιτικής συνοχής, από την χρηματοδότηση κλίμακας, από τη στρατηγική κατάστρωση σχεδίων. Αυτό αλλάζει ωστόσο με τα χρόνια. Κάποιος είπε ότι υπάρχουν στρατηγικές σε, όχι μόνο στην Πολωνία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες που προσπαθούν να θέσουν το πλαίσιο των εθνικών συμφέροντων για την περιφερειακή, τα περιφερειακά ταμεία. Η εθνική ανάπτυξη επίσης προωθείται πιο πολύ και η σύγκληση και όχι τόσο πολύ η περιφερειακή ανάπτυξη και επίσης ε, ε, μία μετάβαση από ένα μοντέλο χαμηλού κόστους σε ένα μοντέλο υψηλής τεχνολογίας, τεχνολογίας ακμής και υψηλού κόστους. Αλλά υπάρχει όλο και πιο πολύ διαφοροποίηση στην ομάδα των χωρών αυτό. Κάποιες χώρες στο κέντρο της Ευρώπης υπερισχύουν σε ό,τι αφορά την απόδοσή τους σε σχέση με χώρες της Ευρώπης των 15. Άρα υπάρχουν διαφορές. Και τέλος, αυτά που ανέφερε ο κ. Τσέλερ για την υποδομή και τις σχετικές δαπάνες στην υποδομή. Εξετάζοντας την ιστορία και το τι γνωρίζουμε για την Ευρώπη των 15, και τα πιο καινούργια κράτη-μέλη. Η... Διαφορές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ποιότητα των δαπανών έχουν να κάνουν με την ικανότητα στρατηγικής ανάλυσης και δικαιολόγησης ε, ανάθεση του κονδυλίου. Υπάρχουν λοιπόν ε, διάφορες ε, υποδομών και λόγω πολιτικών αλλά και λόγω διοικητικών ε, ικανοτήτων, αλλά κυρίως επειδή οι μονάδες γνωρίζουν συγκεκριμένα πράγματα που είναι λιγότερο περιπλοκικά ως μορφή παρέμβασης από άλλες μορφές. Το βασικό θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Τι θα μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μία από τις μεγάλες ευκαιρίες στην επόμενη περίοδο είναι η εξής αν υπάρχει φιλοδοξία για πολιτική με πιο πολλά αποτελέσματα και αν αυτή η πρωτοβουλία και η φιλοδοξία εφαρμοστεί, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, για την υποβολή αναφορών. αναφορών. Που θα καταδεικνύουν με σαφήνεια το τι συμβαίνει επί τόπου. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία να υπάρχει μεγάλη ειλικρίνεια στον εντοπισμό των προβλημάτων. Και ενδεχομένως και αυτή η Επιτροπή εδώ κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει η Επιτροπή Προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά την διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Αλλάζουν οι όροι ξέρετε, αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστούμε, Τζον, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Φρύπτου. Ευχαριστώ. Ακούστηκαν ορισμένα ερωτήματα για την εμπειρία της Ρουμανίας. Την προετοιμασία για την ολοκληρωμένη αστική προσέγγιση. Δύο σχόλια εδώ. Ετοιμάζεται η δημόσια διαβούλευση που είναι πολύ σημαντική για την αστική ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα που δεν θα, που θα αναφέρω λεπτομέρειες αλλά υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες εδώ. Δεύτερον, προετοιμάζονται προγραμματικά έγγραφα εδώ υπάρχει καλύτερο συντονισμό Παραδείγματο χάρη μία παρουσίαση εδώ έλεγε, έλεγε ότι η συμπερίληψη τέτοιων προγραμμάτων στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υπάρχει παντού, αλλά στη Ρουμανία στα περισσότερα υπάρχει. Υπάρχει. Με κύριο στόχο τις λιγότερο προνομιούχες περιοχές και το ίδιο το αστικό περιβάλλον. Και έτσι φύγονται πολλά προβλήματα από, την κοινωνική, από τον κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι πολλά άλλα. Υπάρχει εδώ ανοιχτό πνεύμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Συνοχής, διότι ήδη από τη φάση του σχεδιασμού προσπαθούμε να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν διάφορα προγράμματα διατηρώντας βέβαια τους ισχύοντες κανόνες και το σημαντικότερο είναι ότι από τα πιλωτικά προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα μέχρι τώρα χωρίς να ζητάμε από την κοινωνία των πολιτών, αν δεν ζητήσουμε από την κοινωνία των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση να λύσει τα τοπικά προβλήματα, δεν θα βρούμε ποτέ τη λύση. Διότι πράγματι οι Δήμοι και οι κοινότητες είναι οι μόνοι ικανοί να διαχειριστούν στις επόμενες φάσεις τα προγράμματα και έτσι να υπάρχει και αποτέλεσμα. Όσο για την πολυχρηματοδότηση, λέγω, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένους μηχανισμούς επιλογής. Είναι κάτι που προσπαθούμε να το πετύχουμε και για τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο συνδυασμού, συνδυασμένης ανάπτυξης και της υπαίθρου και του αστικού περιβάλλοντος. Δεν έχουμε βέβαια κανέναν πολύ πολύπλοκο μηχανισμό, αλλά τουλάχιστον κάποιο συνδυασμό. ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Όσο για το, την αλλαγή του συστήματος διαχείρισης, Φαντάζομαι ότι αφορά το θέμα, το ερώτημα δηλαδή της schimba fără uh, cunoștința comisiei care Και η Κομισιόν το παρατηρεί αυτό και το εποπτεύει δημοσιονομικό έλεγχο που προσέχει πάρα πολύ οτιδήποτε γίνεται ως προς αυτό το σύστημα για τις δημόσιες προμήθειες δεν έγινε καμία αλλαγή στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αλλά φαντάζομαι ότι μερικές από τις καινούργιες χώρες μέλη χρειάστηκε να το αντιμετωπίσουν όπως την ερμηνεία ορισμένων πραγμάτων για γιατί υπήρχε διαφορετική ερμηνεία του ποιος ωφελείται, ποιος διαχειρίζεται, ποια είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή κλπ. Ενώ πρόκειται δηλαδή για το ίδιο κείμενο υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Ξαφνικά η Ρουμανία κατάλαβε ότι τέσσερα διαφορετικά μέρη ερμήνευαν διαφορετικά το ίδιο πράγμα. Και αυτό οδήγησε σε μια τρομερή ένταση στη Ρουμανία. Ξέρετε τα έξι προγράμματα για το εξάβιβλος ε, πάγωσαν και ένας ήταν ο λόγος η έλλειψη εμπειρίας εκείνων που ερμήνευαν. Προσπάθησαν να μεταφέρουν σωστά την ομοθεσία αλλά δεν την ερμήνευσαν πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζουμε όταν τελειώσει αυτό να έχουμε πάρει το μάθημα. Και ένα ακόμη σχόλιο, αν και η ερώτηση δεν αφορούσε ακριβώς εμένα. Η χρήση των υποδομών, η επίπτωση ή ο τρόπος με τον ή ο τρόπος λέγω με τον οποίο λειτουργούν τα ευρωπαϊκά μία, Νομίζω ότι η επίπτωσή τους εξαρτάται από τις προτεραιότητές σας. Θέλετε τη μέγιστη δυνατή επίπτωση ή ένα καλύτερο σύστημα που να οδηγεί στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Γιατί μερικά προγράμματα με φιλόδοξο αποτέλεσμα ή στόχο δεν μπορούν να εφαρμοστούν όπως πρέπει λόγω των ισχυών των κανόνων. Και έτσι αναγκάζεται κανείς να τα περικόψει γιατί δεν θέλει να διακινδυνεύσει τη διακοπή του. Ευχαριστούμε κύριε Άλτα Ζόλα. Yes, ε, Ναι. Θα ήθελα δύο σχόλια να κάνω πλεονέκτημα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δεν θέλω να πω ότι παρότι είμαστε μικρή χώρα, έχουμε μια αλφα αποτελεσματικότητα προ προς την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων. Από την άλλη, δεν νομίζουμε ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση, η προσέγγιση κοινοτική ε, υπονομεύονται. Τα έχουμε δοκιμάσει στη χώρα μας χωρίς προβλήματα. Και φαίνεται ότι είναι ωφέλιμο για τους ενδιαφερομένους. Τι είδους λοιπόν προσέγγιση μπορούμε να προτείνουμε στις τοπικές αρχές ώστε να έχουν ένα θεματικό πρόγραμμα και να ξεκινήσουν μία προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αλλά βέβαια αυτό μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα ανάλογα με, την, με το Δήμο ή την κοινότητα. Ε, μπορεί κάποιες χώρες να μην έχουν την ευκαιρία να κάνουν ε, τις, κάποιες πόλεις μπορεί να έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις σχετικές προκηρύξεις, ενώ για κάποιους άλλους μπορεί να είναι το σύστημα ωφέλιμο, χρήσιμο και αποτελεσματικό. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μιλάμε για ε, ό,τι να είναι ή ότι μιλάμε για δαπάνες ε, άκρητα, εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένε δαπάνες. Άρα χρειαζόμαστε αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με, με τις τοπικές αρχές. τώρα στην άλλη ερώτηση, που μερικές φορές δεν είναι αποτελεσματικές. Συμφωνώ απολύτως με τις παρατηρήσεις σας και στις ε, υποδομές όπως τα συστήματα καθαρισμού λιμάτων, διαπιστώσαμε κι εμείς ότι λίγα νοικοκυριά αναλογικά συνδέονται αυτά τα συστήματα. Εκεί και εμείς λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε τις πιο χρήσιμες και αποτελεσματικές λύσεις, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έχουμε κανένα μαγικό ραβδί. Τρεις πιθανές λύσεις έχω να προτείνω. Μία που θα είναι να συζητήσουμε και να εντοπίσουμε ενδεχόμενα προβλήματα. Αφήνοντας και ένα περιθώριο ευελιξίας, γιατί η καταστροφή του 2018 μπορεί να είναι τελείως διαφορετική και πρέπει να αφήσουμε ένα περιθώριο για προσαρμογή όταν έρθει η ώρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Μια άλλη παρατήρηση, εταιρική σχέση. Ξέρουμε ότι έχουν ήδη γίνει συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάλι οι τοπικές αρχές φαίνονται ικανοποιημένε. Και έτσι, εάν ζητήσουμε από τοπικές αρχές, αν ζητήσετε από τοπικές αρχές κοινωνικού εταίρους και με κυβερνικές οργανώσεις να συμμετάσχουν, θα δείτε ότι είναι γενικά καλή εικόνα που δίνεται. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προτείνουμε, τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύουμε ότι έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Μπορεί να επαληθεύει τα προγράμματα της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, της προγραμματιζόμενες δαπάνες. και να αναζητεί αποτελέσματα διευκολύνει την συνεργασία με άλλους εταίρους, την ανάλυση των καταστάσεων και αναγκών ή και πιθανών λύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλεντόφσκι, ευχαριστώ εν συντομία σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία. Πώς ε, γίνεται η εποπτεία. Πολύ σημαντική αφορα την μεθοδολογια πως γινεται η υποπτία. πολυ ότι το scoreboard για την περιφερειακή καινοτομία για την παρακολούθηση της καινοτομίας αυτής ξεκινάει με τους μετριοπαθείς αν θέλετε καινοτόμους. Το πιο σημαντικό όμως είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από τους δείκτες. Τι συμβαίνει πραγματικά. Μπορούμε λοιπόν έτσι να δούμε καλύτερα τις περιφέρειες, τους βασικούς καινοτόμους. και οι περιφερειακές περιοχές, περιφέρειες, με υψηλό επίπεδο απασχόλησης και παραγωγής, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πρόκειται για περιφέρειες που έχουν, για παράδειγμα, γνώση, παρέχουν υπηρεσίες, έχουν πιο λειτουργική προσέγγιση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε, και αυτό είναι σημαντικό, τι συμβαίνει πίσω από τους δείκτες αυτούς. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τις περιφέρειες στη τελική ανάλυση είναι να βρουν συγκεκριμένα αξιόπιστα μέτρα και τον θετικό αντέκτυπο αυτών. Και νομίζω ότι προς τα εκεί οδεύει το νέο πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια της κυρίας Προέδρου, κατά πόσο θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη προετοιμασία προς μια συνεργατική προσέγγιση. Αυτό αρχίζει και συμβαίνει σιγά σιγά. Αν έχει να κάνει με το πολιτισμικό, την πολιτισμική πτυχή του θέματος, αλλάζει η κουλτούρα. Αλλά βασικό είναι να κοιτάξουμε και τις ε, συνθήκες που διαμορφώνουν το πλαίσιο και πώς διαμορφώνονται σε σχέση και με τις εταιρείε. Άρα, θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι να βρούμε η απειλή, αν θέλετε, η πρόκληση είναι τι γίνεται με τις ε, περιοχές εξειδίκευσης να δούμε και να διδαχτούμε από τα διδάγματα της προοπτικής της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου και σε ό,τι αφορά τα κριτήρια που επιλέγονται. Και αυτό ενδεχομένως να αντικαταστήσει αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη που υπάρχει. σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και σε αυτό το μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμενους που ήρθαν εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και η συζήτηση που ακούσαμε και από τους υπουργούς. Σας ευχαριστώ και περνάω γρήγορα γρήγορα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ελπίζω να είναι το πέρα κύριε Βάτερσοτ. Ε, τότε θα κάνουμε την παρουσίαση της ε, έκθεσης της Κομισιόν για την ποιότητα της παιδείας στις διάφορες περιφέρειες. Και υπάρχει και η δήλωση στα μέλη της Επιτροπής Περίφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε βουλευτέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή σας επιλέγει τη Γενική Διεύθυνση για την Παιδεία και τον Πολιτισμό της Κομισιόν να παρουσιάσει αυτήν τη μελέτη που λέγεται Mind the Gap οι ανισότητες στην παιδεία μεταξύ των περιφερειών. Θα σας παρουσιάσω πρώτα τα συμπεράσματα της έκθεσης και μετά μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε για το μέλλον. Έχουμε και αντίτυπα που μπορούμε να μοιράσουμε εδώ στην αίθουσα και φυσικά υπάρχει και στην ιστοσελίδα. Λοιπόν, πρώτον, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν μεγάλες ανισότητες στην παιδεία στις διάφορες περιφέρειες πράγμα που δείχνει και ευρύτερε ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, όχι μόνο στην παιδεία, συνδέεται με θέματα οικονομικής ανάπτυξης και παιδείας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μερικοί πεπαιδευμένοι άνθρωποι να φεύγουν από την περιφέρειά τους λόγω της διαρροής εγκεφάλων διότι μπορεί να είναι εκπαιδευμένοι αλλά φεύγουν παρόλα αυτά και άρα φεύγει και η γνώση από την περιφέρεια. Και αυτό έχει επιπτώσει μετά στη συνέχεια στην οικονομική ανάπτυξη κλπ. Είναι πρόβλημα. Και φυσικά αφορά και θέματα κοινωνικής συνοχής γιατί οι ενισότητες στην παιδεία μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική συνοχή. Ε, e so, a Λοιπόν, αρχίζω με την εκθέση που έχουμε εδώ στα χέρια μας. Υπάρχει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τις κοινωνικές πτυχές της εκπαίδευσης και της παιδείας που αναλαμβάνουν μελέτες για την Κομισιόν. Και εδώ πρόκειται για μία εξέταση γενικά των εμπειρικών δεδομένων που έχουμε για τις ε, ανισότητες στην παιδεία και από το Ευρωστάτ αλλά και από άλλες πηγές όπου υπάρχουν. Η ομάδα αυτή των κοινωνικών επιστημόνων με επικεφαλή τον Δημήτρη Μπάλα και τον κύριο Ντάνι Ντόρλινγκ είχαν προσκληθεί αλλά δεν μπορούν να προσέλθουν είναι πολύ υψηλού επίπεδου ομάδα η εκθέση συμπεριλαμβάνει πάνω από 100 χάρτες που δείχνουν αυτές τις ε, ανισότητες στην παιδεία έχει φυσικά και τα όρια του. Στο, σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2 είναι τα περισσότερα στοιχεία. Πιο λεπτομερή κατανομή δεν έχουμε και γι' αυτό δεν είναι εξαιρετική η σύγκριση που μπορούμε να κάνουμε μεταξύ των χωρών. Εξάλλου υπάρχουν και απαρχαιωμένα στοιχεία από το 10 μερικές φορές. Αλλά όλα αυτά κάτι μας δείχνει. Προσπάθησε η έκθεση αυτή να βασίσει τους χάρτες της σε 12 διαφορετικούς δείκτες που αφορούν τις δυνατότητες εκπαίδευσης και τα άλλα κυριότερα θέματα. Ποια είναι τα βασικά θέματα λοιπόν. Πρώτον, προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα ποιες είναι οι περιοχές που είναι πιο μειονεκτικές ως προς την παιδεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεύτερο ερώτημα. Πώς συγκρίνονται οι χώρες μέλη ως προς την εσωτερική τους κατανομή των ε, εκπαιδευτικών ανισοτήτων μέσα σε κάθε χώρα δηλαδή. Και το τρίτο, τι μέτρα θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα αυτό των ανισοτήτων. Ας δούμε λοιπόν τους χάρτες. Ένας βουλευτής εδώ νομίζω είπε ότι είναι δύσκολο να βλέπει κανείς τις μικρές οθόνες. Καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι δύσκολο να διαβάσετε αυτούς τους χάρτες, αλλά ελπίζω να τους κοιτάξετε και στο δημοσίευμα. Αρχίζουμε με την ανάλυση μεταξύ χωρών. Έχουμε όλο το χάρτη εδώ της Ένωσης. Ο πρώτος δείκτης είναι πόσοι είναι ανειδίκευτοι ή αμόρφωτοι. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι θύλακε, βέβαια περιοχών ανθρώπων που είναι τελείως ανειδικευτοί και αμόρφωτοι, άλλοι που έχουν φτάσει μέχρι το γυμνάσιο και μπορεί κανείς να δει ότι υπάρχει εδώ ένας διαχωρισμός βορρά-νότου. Στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές ανισότητες. ναι, είναι και το Βέλγιο εκεί. Λοιπόν, συγκεκριμένες περιφέρειες. Αυτές που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό ανειδίκευτων είναι το Αλεντέχο στην Πορτογαλία, Θέντρο Πορτογαλία, Νόρτε Πορτογαλία, Εστρεμαδούρα στην Ισπανία κλπ. Ε, αυτές είναι οι χειρότερες περιπτώσεις, ενώ ε, οι περιφέρειες όπου υπάρχουν πολύ λίγοι ανειδικευτοί είναι στην Πράγα και σε γερμανικές περιφέρειες. Τώρα να δούμε πώς κατανέμονται οι ψηλά εκπαιδευμένοι. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Ο χάρτης δείχνει όσους έχουν λάβει ανώτερη εκπαίδευση και διπλώματα. Εδώ δεν υπάρχει συγκέντρωση, δηλαδή ο υψηλότερος αριθμός ανθρώπων με τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται στο Λονδίνο, Μπραμπάν στο Βέλγιο, στο Χόλμη, Βασκία, Οτρέχτη κλπ. Και η περιοχή των Βρυξελών. Και οι περιοχές που υπάρχει πολύ λίγη τριτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο 7% είναι στο Σεβέρο Ζάπαντ στην Τσεχία Σουντ Μοντένια στη Ρωμανία, η Βάλεντα Όστα στην Ιταλία και πάλι το Αλεντέχο στην Πορτογαλία. Υπάρχει κάποιος σχετισμός λοιπόν μεταξύ των δύο χαρτών. Τώρα είδαμε όσους έχουν χαμηλή εκπαίδευση, όσους έχουν υψηλή. Τώρα να δούμε ποιοι συμμετέχουν στη διαβίου μάθηση που είναι και αυτός ένας δείκτης. Εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλες ανισότητες ολόκληρη την Ευρώπη. Ο διαχωρισμός δεν είναι βορράς-νότος, αλλά βορράς-νότιο-ανατολή. Ο υψηλότερος αριθμός συμμετεχόντων στη διαβίου μάθηση είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Δανημαρκία, στη Φιλανδία και τη Σουηδία, ενώ ο χαμηλότερος αριθμός στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Μερικά παραδείγματα, πολύ χαμηλή συμμετοχή στη Βουλγαρία, το Σεβροζαπάντιν, στην Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, στερεά Ελλάδα, Στη Βουλγαρία πάλι Γιουγκολτσλόχεν Σλόχεν και Σέβερο Ιστόχεν. Ενώ ο υψηλότερος αριθμός συμμετοχής είναι σε πολλές πόλεις και περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Λονδίνο, στο Χόβερστάντεν στη Δανία, Μιτ Γιούλτλαντ κλπ. Καθώς και στη Φιλανδία και Σουηδία ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Τώρα τελικά οι ανισότητες μεταξύ περιφερειών και χωρών γεωγραφική πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση. Δείχνει πού ζει ο πληθυσμός σε απόσταση άνω των 60 λεπτών από κάποιο πανεπιστήμιο. Αυτό βέβαια είναι καθαρά γεωγραφικό κριτήριο, αλλά πάλι ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ είναι στη Θέουτα και πάλι στη βουλγαρική περιοχή της Εύερος Μάλτα, Μερία και περιφέρειες της Ελλάδας. Βέβαια κανείς πρέπει να τα όλα αυτά με κάποια προσοχή γιατί υπάρχουν τώρα περισσότερες δυνατότητες διαβίου μαθήσεως ή μέσω ίντερνετ. Επίσης παρατηρούμε ότι ο δείκτης αυτός δεν δείχνει τίποτα θετικό για τη βόρεια, για το βορρά της Ευρώπης, Σουηδία, Φιλανδία. Ενώ από άλλους χάρτες είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη μόρφωση εκεί. Τώρα μεταξύ, μέσα σε κάθε χώρα μέλος μάλλον, ποιο είναι το χάσμα μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων αριθμών πεπαιδευμένων σε μία χώρα. χαμηλός δείκτης η εδώ είναι οι αριθμοί που δείχνουν τις, τα μεγαλύτερα χάσματα χαμηλότερα στην Αλσατία υψηλότερα στην Κορσική αυτό είναι το μεγαλύτερο χάσμα. Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Γερμανία επίσης δείχνουν μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν λίγες ανισότητες σε χώρες όπως η Σλοβενία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Αυστρία και Φιλανδία. Και βέβαια πάλι μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτόν το δίκτυ με κάποια φρόνηση γιατί αν μια περιφέρεια έχει χαμηλό μερίδιο στην μόρφωση και άλλη είναι απλώς καλύτερη χωρίς να είναι άσκημη η οικονομική κατάσταση της άλλης περιοχής πάλι θα βρεθεί χειρότερη στον Τώρα, φοιτητέ σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μάλλον για το μέλλον, γιατί είναι φοιτητέ που είναι εγγεγραμμένοι τώρα. Και αυτό θα δείξει στο μέλλον ότι θα μετρηθούν μεταξύ των πεπαιδευμένων. Εδώ φαίνεται, φαίνονται πάλι τεράστιες διαφορές που οφείλονται στην ύπαρξη περισσότερων πανεπιστημίων στις πρωτεύουσες. Το μεγαλύτερο χάσμα είναι μεταξύ Βρυξελών και περιφερίας του Λουξεμβούργου του Βελγίου. Επίσης μεγάλα χάσματα στην Τσεχία, Αυστρία και Ιταλία. Η Ελλάδα και η Ρουμανία επίσης έχουν χάσματα άνω του 80%. Αλλά βέβαια αυτό εξηγείται συνήθως από το γεγονός ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται περισσότερο στις μεγάλες πόλεις ή τις πρωτεύουσες. Τώρα κάτι, πιο, κάτι λίγο διαφορετικό. Η πραγματική φίτηση των φοιτητών. Εδώ βλέπουμε μια λίγο διαφορετική εικόνα και κατάλογο χωρών. οι αποφυτούντες, οι απόφοιτοι και εδώ υπάρχουν μεγάλα χάσματα μεταξύ περιφερειών στην κάθε χώρα. Φοιτητών που δεν έχουν αποφοιτήσει δηλαδή και φοιτητών που έχουν αποφοιτήσει. Μεγάλα χάσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Τσεχία, Ισπανία, Σλοβακία, Ρουμανία. Πάλι οι ίδιες περιφέρειες εμφαίνονται στη Γαλλία, 33% γύρω από την πρωτεύουσα, ενώ στην Κορσική μόνο 11%. Επίσης όπου είναι μικρά τα χάσματα, που στην Ιρλανδία, Ιταλία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Φιλανδία και Αυστρία, κάτω του 10%. Και τελευταίος δείκτης πάλι για τις ανισότητες μέσα σε κάθε χώρα μέλος, συμμετοχή των ενηλίκων στη διαβίου μάθηση. Μεγάλο χάσμα για το Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβακία και Δανία, αλλά αυτό εξηγείται από το ότι ήδη έχουν πολύ υψηλή συμμετοχή στη διαβίου μάθηση ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι υπάρχει ένα θέμα ανισότητας εδώ. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Υπάρχουν πολύ περισσότερα στοιχεία βέβαια από όσα σας παρουσίασα. Αν ενδιαφέρεστε διαβάστε το έγγραφο. Αλλά να σας πω τώρα μερικές σκέψεις για την πιθανή λήψη μέτρων μπορεί να σας ενδιαφέρει. Η μελέτη δείχνει ότι το που ζει κανείς στην Ευρώπη επηρεάζει το μορφωτικό του επίπεδο και άρα και τις επαγγελματικές του προοπτικές. Σημαντικό συμπέρασμα αυτό. Επίσης πρέπει να ξέρουμε, αν και ίσως δεν είναι αυτή η καταλληλότερη επιτροπή, Οι εθνικοί μέση όροι καμιά φορά βέβαια κρύβουν τις ανισότητες περιφερειακές, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί να ενδιαφέρει και την Επιτροπή σας το θέμα των ανισοτήτων. Τι μπορεί να κάνει κανείς λοιπόν. Δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που έχουν ήδη εφαρμοστεί και πολλές φορές έχουν κάνει προσπάθειες για να μειώσουν τα χάσματα, αλλά αυτό που μπορούμε να πάρουμε ως μάθημα είναι ότι οι χώρες έχουν μία, ένα προσέγγιση ανακατανομής των κονδυλίων μεταξύ περιφερειών ή εφαρμόζουν πιο στοχευμένα προγράμματα σε συγκεκριμένες περιφέρειες Υπάρχουν τέτοια προγράμματα στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Σουηδία κλπ. Εξαρτάται λοιπόν από τις ανάγκες της κάθε περιοχής η στοχευμένη προσέγγιση. Άλλο όμως πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ανάγκη να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα της παιδείας χωρίς να το συνδέσουμε με άλλα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της ίδιας περιφέρειας. Σας το έλεγα και στην αρχή, οι ανισότητες μεταξύ περιφερειών συνδέονται πολλές φορές με το εισόδημα, με την οικονομική ανάπτυξη, με την απασχόληση. Οποιαδήποτε μέτρο λοιπόν πρέπει να έχει και τέτοιο εύρος. Όχι να περιορίζεται μόνο στην παιδεία καθεαυτήν. Τέλος. Ίσως το σημαντικότερο δίδαγμα είναι ότι όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν τη σημασία που έχει το ανθρώπινο κεπάλαιο που είναι ένας από τους παράγοντες για την περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό. Όπου υπάρχει γνώση, ελκύει καινοτομία, έρευνα και τελικά ανάπτυξη. Οι οικονομικοί παράγοντες λοιπόν εξαρτώνται από τους ανθρωπίνους τους. Αυτό φυσικά επιβεβαιώνει ότι αξίζει τον κόπο να διευρυνθεί η συμμετοχή στην ανώτερη παιδεία. Αυτό είναι το κύριο δίδαγμα. Και τώρα πώς μπορεί να συμβάλλει η Ένωση. Πολλά μπορεί να γίνουν εθνικά και περιφερειακά, αλλά τι θα μπορούσε να κάνει η Ένωση. Πρώτον, πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Ευρώπη 2020 η στρατηγική αυτή με τους στόχους της για έξυπνη, βιώσιμη και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμό είναι σημαντικό καθώς και η εκπαιδευτική στόχη του 2020 από όπου βλέπουμε ότι και περιφερειακά πρέπει να το δούμε αυτό και άλλο πολύ σημαντικό είναι σαν καθοδηγητικό μέτρο ότι τα τελευταία χρόνια έχει όντως μεγάλη σημασία στο θέμα της παιδείας. Ως προς το επίπεδο εκπαιδευτικής συνεργασίας στην Ευρώπη Υπάρχει η λεγόμενη ανοιχτή μέθοδος για συνεργασία μεταξύ χωρών για την ενθάρρυνση της αμοιβαίας μάθησης και αυτό φυσικά θα συνεχίσουμε να το προσέχουμε και να το ενδυναμώνουμε μάλιστα για να δούμε πώς θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και ισότητα. Και βέβαια και δύο πρόσφατες πρωτοβουλίες. το περασμένο Νοέμβριο η Κομισιόν έκανε μια δήλωση που λέγεται Rethinking Education όπου έλεγε ότι είναι βασικό να αυξηθεί το βαθμός εκπαίδευσης για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, οι δημογραφικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση και ιδιαίτερα τα προσόντα ΒΕΤ που βασίζονται στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επίσης υπάρχει η πρωτοβουλία Opening Up Education που θα την παρουσιάσει αύριο η Κομισιόν. Είναι μια ευρεία, ευρεία, ευρεία σημασίας δήλωση για την ε, μάθηση εξ μέσω ίντερνετ για τις πιο αδύναμες και μη προνομίχες ομάδες. Και βέβαια πρέπει να διευρυνθεί η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αύριο κοιτάξτε την αυτή την ανακοίνωση. Τώρα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, άλλο πολύ σημαντικό. Ο έρασμος συν 14 με 20 θα δώσει περαιτέρω ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνεργασίας συμμαχιών, εκπαιδευτικών οργανισμών, κοινωνικών εταίρων κλπ. με τον αυξημένο του προϋπολογισμό. Και να σας πω και δύο λόγια για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά επενδυτικά ταμεία. Η επένδυση στην παιδεία και την εκπαίδευση, από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, σε συνδυασμό με την συνοχή, δείχνει ότι η επένδυση στην παιδεία είναι ο μόνος τομέας όπου υπάρχουν αποτελέσματα μέσω και μακροπρόθεσμα. Είναι μια πρόσφατη μελέτη που δείχνει ότι μεγαλύτερο, περισσότερο ανθρώπινο κεφάλαιο σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα στις περιφέρειες και μείωση των ανισοτήτων ή μάλλον το αντίθετο ότι περισσότερες ανισότητες σημαίνουν και περισσότε... ε, ανθρώπινες, στο ανθρώπινο κεφάλαιο σημαίνουν και περισσότερες οικονομικές ανισότητες και ότι η τριτοβάθμια και περισσοτερες στο ανθρωπινο οδηγεί συνήθως σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Τώρα τα συμπεράσματα για την πολιτική συναχής. Υπάρχουν ακόμα οι διαπραγματεύσεις βέβαια για το Πολδίπ μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει μεγάλη επένδυση με τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ευρωπαϊκά ταμεία και επίσης αυτό είναι σημαντικό και για το κοινωνικό ταμείο Αυτό το έχουμε λάβει δεόντως υπόψη μας και εμείς. Και για το Περιφερειακό Ταμείο και τις υποδομές της παιδείας. Όταν μιλάμε για το κοινωνικό ταμείο πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να διασφαλιστεί επαρκής επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ό,τι και να κάνουμε βέβαια πρέπει να είναι προσέγγιση που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και με συνεργασία το, με άλλους στόχους η παιδεία μαζί με καινοτομία, έρευνα, απασχολησιμότητα, κοινωνικό, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και με διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι μόνο τον έρασμο αλλά και τον ορίζοντα 2020. Εμείς συνεργαζόμαστε άμεσα με Υπουργεία Παιδείας για να είναι βέβαιο ότι θα συνεννοηθούν με τους αρμόδιους υπουργούς και όταν επεξεργαζόμαστε τα προγράμματα το προσέχουμε αυτό. Uh, basically what I wanted to present. I hope I have not been. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Ελπίζω να σας ενδιέφερε. Ευχαριστώ. Thank you uh, very much. Σας ευχαριστώ θερμά. Βίκτορ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την συμβουλή. Υπάρχουν κάποια, κράτη, κάποια θέματα που είναι σχετικά όχι για κάποιο κράτος μέλος, αλλά για την Ένωση. Κοιτάξτε, καταρχάς, είναι δεδομένο ότι σε πολλά από τα κράτη μας ο αναλφαβητισμός εντείνεται μόνο, αυξάνεται μόνο. Αντίθετα από ό,τι έχει συμβεί σε προηγούμενες κρίσεις. Αυξάνεται διαρκώ ο αναλφαβητισμό. Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για εκπαίδευση όταν έχουμε φαινόμενο μαζικού αναλφαβητισμού. Δεύτερον, εντυνόμενη τάση και το, η αύξηση του χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. Και αυτό δεν χαρακτηρίζει μόνο τη δική μου χώρα ή τη Βουλγαρία. Επίσης, αυξάνονται τα χάσματα μεταξύ των πανεπιστημίων mm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν εξαιρετικά πανεπιστήμια, αλλά υπάρχουν και πανεπιστήμια τα οποία δεν μπορούν καν να αναχθούν στο επίπεδο των εθνικών προδιαγραφών που έχουν ορίσει. Επίσης, όταν ένας ε, εξαίρετος φοιτής, ένας λαμπρός φοιτής έχει πάρει το πτυχίο του και μένει άνεργος, τι έχουμε να του προσφέρουμε εμείς. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ισπανία. Όλες οι χώρες έχουν πρόβλημα ανεργίας των νέων και όλες οι κοινωνίες καλούνται να δώσουν μια απάντηση. Πώς θα πείσουν τον νέο να πάει στο πανεπιστήμιο σε μια πολύ ασταθή αγορά εργασίας. Εκεί όταν το μέλημά του είναι μόνο να βρει μια θέση εργασίας και λιγότερο καλά αμοιβόμενη και με λιγότερες απαιτήσει. Απλώς να είναι μια δουλειά. Και αυτό στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ ξεκάθαρο. Στην ε, Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, δεν ξέρω αν και η Πολωνία έχει το ίδιο φαινόμενο. Οι νέοι μα φεύγουν, ψάχνουν καλύτερε θέσει εργασία στην αγορά τη Ευρώπη. Πράγμα το οποίο είναι φυσιολογικό γιατί αυτό επιβάλλει η φιλοσοφία της αγοράς. Αλλά ποιος θα μείνει τελικά να ηγηθεί των κοινωνιών μας, των τοπικών αρχών, Εδώ έχουμε να κάνουμε με τραγικά, τραγικών επιπτώσεων ερωτήματα. Η Κίνα πρέπει να σας πω είναι στη θέση να προσφέρει θέσεις εργασίας για 5 εκατομμύρια φοιτητές ε, με το που παίρνουν το πτυχίο τους δηλαδή έχουν προσληφθεί. Ξέρω ότι έχουμε διαφορετικά μεγέθη. Αλλά το ένα, η μία εικόνα μας δείχνει ε, εργαζομένους με υψηλή κατάρτιση και από την άλλη έχουμε μια γενιά υψηλής κατάρτισης που δεν βλέπουν θέσεις εργασίας του από το μικροσκόπιο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ένα ερώτημα που αντιμετώπισε και ο Μάρτιν Σούλτ στην ε, συνάντηση που είχε με τους φοιτητέ. Επομένως, ή θα πρέπει να φεύγουν οι νέοι σε διάφορες χώρες, γιατί δεν μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας. Ή θα πρέπει να δώσουμε τη λύση για την απασχόληση μιας νέας γενιάς με πολύ πολλές δεξιότητες. Ευχαριστώ πολύ, Βίκτορ. Πρέπει να τελειώνουμε όμως. Ο κύριος Όλριχτ. Ναι, ξέρω ότι έχουμε μείνει και λίγοι, αλλά να κάτσουμε και λίγο παραπάνω, γιατί όχι. Εγώ κοιτάω τα αποτελέσματα και τα δεδομένα. Και μια ερώτηση είναι αφού εντοπίζονται οι αποκλήσεις και οι Έλληνες τι οφείλονται. Φταίει το επίπεδο τη κατάρτιση, τη ε, ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, τη ύπαρξη σχολείων, τι από όλα αυτά. Γιατί οι διαφορές οι αποκλήσεις είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή βλέπουμε διαφορά σε σχέση με την ε, επαρχία Λουξεμβούργου του Βελγίου, η οποία έχει πολύ χαμηλό επίπεδο. Ε, δεν θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Αυτό νομίζω θα πρέπει να κοιτάξουμε. Θα είμαι σύντομη κι εγώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με το όσο είπε ο Γιάννο Ολβρίχτ. Ευχαριστώ την ομιλήτρια. Θα συστήσουμε λοιπόν αυτό που μας παρουσιάσετε για τα μία συνοχής και τη χρήση τους. Ο στόχος φαντάζομαι της παρουσίες ήταν τα μέτρα, η εξέβρεση των μέτρων που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Πολύ ωραία, υπόθηκε αυτό. Αλλά πώς θα λύνουμε το θέμα και ποια μέσα έχουμε σε θέση μας. Έχουμε λοιπόν κάποια μέσα, το ξέρουμε πολύ καλά. Πώς αξιοποιούνται όμως και τι είδους αποτέλεσμα μπορούν να φέρουν ως προς τη μείωση αυτών των ε, αποκλήσεων. Αυτό διότι αφού άκουσα τα όσα είχατε να πείτε και εσείς και οι ομιλητές όλοι, ε, διαρωτώ με τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. ή πού μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί από τη μια επιτροπή στην άλλη μας παρουσιάζονται διάφορε εκθέσεις. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή όμω αυτές όλες να τις διασταυρώσουμε για να δούμε πού βρίσκονται τα καλύτερα παραδείγματα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είμαστε πιο ε, να, να, να δίνουμε πιο αυστηρές οδηγίες για τη χρήση των κονδυλίων. Ίσως και αυτό είναι μια λύση. Μια σειρά από ερωτήματα λοιπόν. Αν τα είχαμε ακούσει όλα αυτά πριν από κανένα χρόνο, μπορεί να είχαμε διαφορετική αντίληψη και αποφάσεις. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά έχετε δύο λεπτά μόνο στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Ίσως μπορείτε να αλλάξετε ύστερα και συνδέσμους με τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται. Ναι, ναι, ναι, φυσικά να συζητήσουμε και μετά από τη συνάντηση. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Κατά σειρά. Τα συμπεράσματα αυτά ίσως να έχουν, κάνει, ίσως να έχουν με άλλα ζητήματα. Αλλά ασφαλώς μας μας ενδιαφέρουν πάρα πολλά θέματα. Και έχουμε συγκεκριμένε δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αναλφαβητισμού έχουμε ορόσημα, το κοιτάμε αυτό και σε επίπεδο υψηλού, σε ομάδες υψηλού επίπεδου. Δεν έχουμε πατρελαιτητά όμω τα περιφερειακά τέτοια στοιχεία και αυτό αποτελεί ένα θέμα στην όλη χαρτογράφηση. Το θέμα τη ανεργία μετά την αποφύτιση. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα θέμα που πλήττει ιδιαίτερα σε κάποιες χώρες. τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνουμε ότι ότι όσο πιο πολύ εκπαίδευση έχει ένα άτομο, τόσο λιγότερη πιθανότητα έχει να καταλήξει άνεργος. Άρα είναι η καλή επένδυση, ακόμα και αν τελικά δεν βρει δουλειά κατευθείαν μετά την αποφύτιση. Για την, ε, το brain drain. Έτσι είναι τα πράγματα όπως λέτε. Δεν υπάρχει ούτε κάποια μυστική, ούτε κάποια μαγική λύση. Είναι ένα ευρέω δεδομένο φαινόμενο που έχει να κάνει με την περιφερειακή ανάπτυξη. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται επένδυση σε ικανότητε και αυτό ασφαλώ θα προσελκύσει οικονομική δραστηριότητα στι περιφέρειες. Ποιοι είναι οι λόγοι που υπάρχουν διαφορέ και τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μα. Βρισκόμαστε στην επαρχή της διαδικασία γιατί η μελέτη ήταν πολύ χαμηλού προϋπολογισμού. Νομίζω ότι ξοδέψαμε λιγότερο από 8.000 ευρώ σε αυτή τη χαρτογράφηση. Ουσιαστικά δηλαδή απλά ε, δένουμε μαζί ήδη υφιστάμενες πληροφορίες. Έχουμε σχετικές εργαλεία, σχετικά εργαλεία, γνωρίζοντας φυσικά ότι πρόκειται για εθνικές αρμοδιότητες. Έχουμε κάποια εργαλεία πολιτικής, έχουμε ασφαλώς ε, μια μεγάλη δυνατότητα επενδύσεων στα ερευνητικά ταμεία και τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να γίνει αυτό. Να δούμε και τι γίνεται να γίνει παραπάνω έρευνα σε βάθος χρόνου. Αφετέρου, αυτά που κάνουμε τώρα είναι το εξής. Αναλύουμε υπηρεσίες μας έχουν αναλυτές αναχώρα και εξετάζουμε τι γίνεται αναπεριφέρεια, αναχώρα, ποιες είναι οι προκλήσεις στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, προκειμένου να υπάρξει ένα... μια συμφωνία σχετικά με τις προτεραιότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Λαϊκή Πρόεδρος. Ελπίζω όταν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να γίνει μια συνέχεια της μελέτης, να μας παρουσιαστεί γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έκθεση της συνεδρίασης των συντονιστών έγιναν σημαντικές αποφάσεις, Ε, Δώσαμε στο ΕΛΚ ε, την έκθεση για το Ταμείο Αλληλεγγύης το Συμβούλιο του Ιουνίου οδήγησε σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοοικονομική εκχώρηση τέτοιων κρατών μελών και αυτή στο ΕΛΚ για την βιολογική βιομηχανία στο ΕΛΚ τις γαλλικές περιοχές εξοχώς αποκεντρωμένες στους σοσιαλιστές για τις Κανάριες νήσους στο ΕΛΚ μέτρα για την Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά Ηλεκτρονικής ε, Επικοινωνίας ε, στους πράσινους. Λάβαμε αποφάσεις για τις αντιπροσωπείες. Υπάρχει μια πρόταση για αντιπροσωπεία στην Ολλανδία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε λάβει ακόμα προτάσεις σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην αποστολή αυτή. Όσοι ενδιαφέρονται τα αρχιστά παρακαλώ να μιλήσουμε τους συντονιστές. για το επόμενο έτος, τους τρεις μήνες μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, μπορεί να υπάρξει μια άλλη αντιπροσωπεία και άλλη μια ακρόαση τουλάχιστον. Θα συναντηθούμε με τους συντονιστές, θα μας δώσουν τις πληροφορίες μέχρι τις 11 Οκτωβρίου και μετά αποφασίσαμε για να γίνει και μια εξωτερική μελέτη η οποία ελπίζω να ενδιαφέρει και το νέο κοινοβούλιο για την πολιτική συνοχή 2014-2020 αποφασίσαμε επίσης να προσθέσουμε στην ήδη υφιστάμενη μελέτη για την ετοιμότητα των κρατών μελών για τη νέα πολιτική συνοχή στο θέμα της αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας των κρατών μελών και άλλο ένα θέμα να σας πω. Χωρίσαμε διαγνωμοτοτήσει για προτάσει οδηγία και προτάσει κανονισμού σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος του Μαγιότ ο κύριος Τριουλιέν θα ήταν ο εισηγητή. Τώρα πλέον ενημερωθήκαμε ότι οι δύο επιτροπέ η και θα τα εγκρίνουν τον ε, Νοέμβριο και θα πάει στα Λομέλια τον Δεκέμβριο και άρα θα ανοίξει τώρα η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και μετά οι τροπολογίες 14 Οκτωβρίου θα ψηφιστούν και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα αποτελέσει τη γνωμοδότηση, την τοποθέτηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτή μόνο την διαδικασία μπορούμε να ακολουθήσουμε. Θα σας αποστείλουμε τις πληροφορίες. Επόμενη συνεδρία στις 14 Οκτωβρίου 2013. Πέρας συνεδρία